colleagues, can we, um, can we take our seats so we can uh, start today? Συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ για να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Good. Well, good morning. Good afternoon, everybody. Um, Συνάδελφοι, καλησπέρα σα. Η αντιπρόεδρο Κόμη θα προεδρεύσει για την απογευματινή συνεδρίαση. Θα της παραδώσω την προεδρία σε λίγο. Απλώ πρέπει να κάνω κάποιε ανακοινώσει. Καταρχήν, με μεγάλη μου χαρά, καλωσορίζω τον Μισελ Μπαριέ, που όπω γνωρίζετε είναι υποψήφιο επίτροπο για την εσωτερική αγορά και τις υπηρεσίε. Συγχαρητήρια Ήσασταν πολύ δραστήριο μέλος της Επιτροπής μας και προσβλέπουμε ε, σε μια μελλοντική συνεδρίαση της Επιτροπής θα κάθεστε εδώ μπροστά μας όπου θα σας ε, υποβάλουμε εμείς τις ερωτήσεις. Χαρά μας λοιπόν που είστε εδώ σήμερα. Δύο, παρα... δύο σύντομε ανακοινώσει. Καταρχήν, η επικοδομητική συνεδρία των συντονιστών μόλι ολοκληρώθηκε. Διάφορα σχέδια μα απασχολούν. Θα σα τα αναφέρουμε μετά τα Χριστούγεννα. Ε, ιδιαίτερα όσον αφορά κάποιε γνωμοδοτήσει για διάφορε εκθέσει πρωτοβουλία από άλλε επιτροπέ. Οι συντονιστέ θα συζητήσουν με τα μέλη για την ε, ε, κατανομή των γνωμοδοτήσεων και θα επανέλθουμε. Έχουμε επίση πρόταση για προφορική ερώτηση για το δύσκολο θέμα των δανείων για τι ΜΜΕ και θα πρέπει να το συζητήσουμε πριν να μπει στην Ολομέλη. Να σας πω επίσης ότι υπάρχουν δύο προφορικές ερωτήσεις τις οποίες συμφωνήσαμε παλιότερα. Η μία αφορά τα θέματα της χαρτοπεξίας, ε, των τυχερών παιχνιδιών και το άλλο είναι αμοιβές, ε, ε, αμοιβαία αναγνώριση πτυχίων. Πέμπτη πρωί για την επόμενη σύνοδο του Στρασβούργου που θα είναι στις 17 Δεκεμβρίου δηλαδή. Παρακαλώ να είστε παρόντες. Αυτό σημαίνει ότι γι' αυτό και εγκαταλείψαμε δυστυχώς το σχέδιό μας να έχουμε μια νέα συνεδρίαση με τους υπουργού της Σουηδίας ε, την Πέμπτη πρωί, γιατί σαφώς δεν γίνονται και τα δυο ταυτόχρονα. Ωστόσο έχουμε ε, μια άλλη ατραξιόν που είναι στις 6.30 το απόγευμα της Δευτέρας μέχρι τις 8 ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής, όπου ολόκληρη η Επιτροπή θα έχει την ευκαιρία να ακούσει και να υποβάλει ερωτήσεις στον καθηγητή Μάριο Μόντι, που όπως γνωρίζετε ανέλαβε την ειδική μελέτη της Επιτροπής για το θέμα της ε, ε, της εσωτερικής αγοράς. Ελπίζουμε ότι θα είναι παρόν και ο υποψήφιος Επίτροπος Μπαρνιέ και άλλα μέλη της Επιτροπής. 6.30 λοιπόν η ώρα το απόγευμα την Δευτέρα. Αυτές είναι οι ανακοινώσεις μου. Θα δώσω τώρα την Προεδρία στη Λάουρα Κόμη για την υπόλοιπη συνεδρίαση. Ναι, ε, grazie ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα πρέπει εκ των προτέρων να ζητήσω συγγνώμη αν κάνω κάποιο λάθος στα ονόματα. Στα ονόματά σας θα προσπαθήσω να είμαι σωστή. Και σας παρακαλώ να με διορθώνετε αν διαπιστώσετε ότι λέω λάθος τα ονόματά σας. Θα ξεκινήσω άμεσα δίνοντας το λόγο στην κυρία Τούνο, την εισηγήτρια που θα μας ενημερώσει για τη θέση της, για τις τροπολογίες που έχουν υποβληθεί σε σχέση με την έκθεση για το πλαίσιο αξιολόγηση εσωτερική αγοράς και άρα τις τροπολογίες που συνδέονται με την ε, έκθεση της. Και της δίνω το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Για την έκθεση αυτή συζητήσαμε την περασμένη φορά και έλαβα 36 τροπολογίες. Μετά από συζήτηση και ε, μπορώ να δεχτώ τι περισσότερες τροπολογίες, πράγμα που με χαρά σας ανακοινώνω. Στις περισσότερες περιπτώσεις ε, συμφωνώ. Και έχουμε τώρα ένα έγγραφο το οποίο είναι έτοιμο για να ψηφιστεί. Με όλες αυτές τις τροπολογίες που έχετε μπροστά σας. Ορισμένε τροπολογίες αποσύρθηκαν μετά από συζήτηση και έχουμε και τρεις συμβιβαστικέ τροπολογίες που νομίζω ότι έχουν πολύ καλό αντίκτυπο στα έγγραφα της Κομισιόν το καθεστούν δηλαδή πιο σαφές και δίνουν μια προοπτική βελτίωση της κατάστασης της ε, ενίας αγοράς. Νομίζω ότι μετά από όλη αυτή την εργασία από πλευρά μου και από πλευρά των σχεδόν εισηγητών, καθώ και με όσου ε, ενεργά συμμετείχαν και προσέθεσαν τι ιδέες τους υπό τη μορφή τροπολογιών, έχουμε τώρα μια πολύ σαφή πρόταση για βελτίωση της κατάστασης για την μεταγραφή της οδηγίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις όπως αυτή για τις υπηρεσίες στην homepage και για το φόρουμ της εσωτερικής αγοράς, όπου η Κομισιόν με τη δική μας συμμετοχή θα πρέπει να εφαρμόσει. Αν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, είμαι στη διάθεσή σας. Και αν όχι, ίσως οι σκιώδεις ηγητές δεν να πάρουν το λόγο. Ναι, σας ευχαριστώ για την εργασία σας και για την πολύ ε, αποτελεσματική σας παρέμβαση και τώρα θα δώσω το λόγο στους σκιώδες συζητητές και ζητώ συγγνώμη αν δεν το προφέρω σωστά. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Wang Nong. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και την ομάδα της για την εργασία της, γιατί η συνεργασία με τους κοιόδες εισηγητές ήταν ιδιαίτερα καλή και αποτελεσματική σε αυτό το θέμα. Όπως είδατε, έχω καταθέσει διάφορες τροπολογίες που στόχο έχουν να επιμείνω σε τρεις κύριες ιδέες. Πρώτον, η ανάγκη η οθέτηση στο πλαίσιο της υλοποίηση του πίνακα βαθμολογίας για την εσωτερική αγορά, μια πιο ποιοτική προσέγγιση που επιτρέπει να εντοπίσουμε του, τα αίτια της ε, υστέρησης στη μεταγραφή. Το γεγονός ότι αυτός ο πίνακας δεν θα πρέπει μόνο να αποτελεί μέσο πίεσης για τα κράτη-μέλη αλλά ένα εργαλείο κυρίως που στόχο θα έχει να κατανοήσουμε καλύτερα τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη στο πλαίσιο της ε, διαδικασίας μεταγραφής Γνωρίζουμε όλοι ότι η στέρηση στη μεταγραφή μπορεί κάποιες φορές να οφείλεται όχι στην κακή βούληση των κρατών, αλλά στην κακή ποιότητα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που πρέπει να μεταγραφεί. Κατά τρίτο λόγο, υπάρχει ανάγκη να γίνουν περισσότερε προσπάθειε κατά τη διάρκεια τη περίοδου μεταγραφή για να προληφθεί ο κίνδυνο μη μεταγραφή ή εσφαλμένη μεταγραφή, ιδιαίτερα ενισχύοντα τον διάλογο και τι ανταλλαγέ πληροφοριών ανάμεσα στην Κομισιόν και τα κράτη-μέλη. Γνωρίζω ότι η κυρία Τούν συμφωνεί μαζί μου σε αυτά τα διάφορα σημεία και χαίρομαι γι' αυτό. Σε σχέση με τις τροπολογίες που κατέθεσαν τα άλλα μέλη της Επιτροπής ΣΥΜΚΟ, η μόνη πραγματικά προβληματική για την ομάδα μας είναι η παρθόν 19 του κυρίου Χάρμπορ έχω την εντύπωση ότι αυτό το σχέδιο έκθεση για τον πίνακα βαθμολογία τη εσωτερική αγορά δεν είναι το σωστό πλαίσιο για να συζητήσουμε για αυτό το θέμα που γνωρίζουμε όλοι ότι είναι πολύ ευαίσθητο και ελπίζω πω θα μπορέσουμε να το ξανασυζητήσουμε και να βρούμε μια λύση για αυτό το σημείο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Χάρμπορ είναι επίσης και ο δισηγητής. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ κατέθεσα τις περισσότερες τοπολογίες εξ ονόματος ομάδας ε, και του κύριου Βίλαν. Θέλω να σχολιάσω κάποιες από αυτές, ιδιαίτερα θέλω να σχολιάσω αυτή την τροπολογία που κατέθεσα για την δοκιμή της εσωτερικής αγοράς. Είναι τροπολογία 19. Δεν είναι νέα αντίληψη. Είναι κάτι το οποίο έχει ψηφίσει στην προηγούμενη θητεία η Επιτροπή. Και επίσης η ιδέα αυτή βασικά υιοθετήθηκε από την Επιτροπή σε μια από τις προηγούμενες μελέτες που έχουν ε, να κάνουν με το μέλλον της εσωτερικής αγοράς. Εν μέρη, το θέμα που έχουμε είναι ότι υπάρχουν πολλές προτάσεις που προέρχονται από άλλα τμήματα της Επιτροπής και που ενώ μπορεί να ωφελούν ας πούμε, τα, σε θέματα περιβάλλοντος, πολλές φορές οδηγούν στον κατακαιρματισμό της εσωτερικής αγοράς. Και κάποιες αλλαγές σε αυτές τις προτάσεις θα, καθιστούσαν, θα τις καθιστούσαν πιο φιλικές προς την εσωτερική αγορά, χωρίς να υποβαθμίζουν το στόχο τους για την αντιμετώπιση κοινωνικών ή περιβαλλοντικών ή άλλων θεμάτων. Και ακριβώς αυτό προσπαθούσα να κάνω, διότι θεωρώ ότι η είναι βασική ανάγκη να διατηρηθούν οι κύριες αρχές της, της συνθήκης, δηλαδή βελτίωση της εσωτερικής αγοράς, με στόχο την καλύτερη νομοθεσία. Και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να υποστηρίξουμε. Και ελπίζω πως η Επιτροπή θα το υποστηρίξει επίσης. Κάτι ακόμα στο οποίο ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας προέκυψε από τις συζητήσεις που είχαμε με την Κάθριν Ντέι, τη Γενική Γραμματέα ε, της Επιτροπής, και ορισμένοι συντονιστέ ήταν επίσης εκεί. Και Εξετάσαμε και αναλύσαμε τον αριθμό των περιπτώσεων ε, κατά παράβαση που σχετίζονταν με συγκεκριμένες νομοθεσίες για την ενιαία αγορά. Γιατί πιστεύω πως είναι σημαντικοί δείκτες αυτοί για το ποιες νομοθεσίες δημιουργούν, προκαλούν μάλλον προβλήματα, είτε στη μεταγραφή από τα κρατημέλη, είτε αβεβαιότητα λόγω της περιπλοκότητάς τους. Νομίζω λοιπόν πως μια λογική χρήση του πίνακα βαθμολογίας της εσωτερικής αγοράς θα πρέπει να μας δώσει και δείξει και έναν ε, τρόπο ε, για το πώς θα πρέπει να προχωρήσει η εσωτερική αγορά και η νομοθεσία της. Αυτά ήθελα να τονίσω και να ευχαριστήσω κυρίως την εισηγήτρια για τον επικοδομητικό τρόπο με τον οποίο συνεργάστηκαν ε, τα γραφεία μας. Και να την ευχαριστήσω γιατί συμφωνεί με τις περισσότερες από τις τροπολογίες μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στην κυρία Ρούλε. Ευχαριστώ. Κύριε Χάρμπορκ, ε, συμφωνώ με την τροπολογία σας 28 που θεωρώ ότι είναι εξαιρετική γιατί οι διαδικασίες παραβιάσεως είναι εξαιρετικές αν η νομοθεσία δεν ακολουθεί την πορεία που έπρεπε να ακολουθήσει. Εγώ παραδείγματο χάρη πάντοτε κοιτάω για να δω πού υπάρχουν προβλήματα και γι' αυτό καλό είναι να αναφέρετε. Έχω διαφορετική άποψη για την τροπολογία σας 19 διότι αν ε, την κοιτάξουμε από κοντά, σήμερα ξεκινάει η ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας, όπου λέγεται σαφώς ότι η εσωτερική αγορά έχει και οικολογικούς και κοινωνικούς στόχους. Οπότε η διατύπωση του ισορροπολογίας 19 ε, είναι τέτοια ώστε δεν μπορώ να την επικροτήσω. Και έχω μία τελευταία παρατήρηση που αναφέρεται στους χιώδεις εισηγητές των σοσιαλιστών και έχω προβλήματα με την τροπολογία 1 διότι είμαι υπεύθυνη για τις δημόσιες προμήθειες και όταν διαβάζω ότι πρέπει κανείς να αγοράζει τα φθηνότερα υλικά και προϊόντα βρίσκω δεν είναι σωστό όχι με τις χαμηλότερες τιμές είναι κάτι το, με το οποίο δεν μπορώ να συμφωνήσω. Ευχαριστώ και τώρα δίνω το λόγο στον Δόκτωρα Λόγκαρντ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα εδώ να σχολιάσω καταρχήν την παράγραφο 4α διότι προτείνω να προσθέσουμε στο θέμα αυτό των, ε, ε, ομάδων εργασίας In order to σε επίπεδο ομάδα εργασίας αλλά και γενικότερης ε, ε, παρακολουθήσεως να ε, έχουμε υπόψη μας ότι εδώ συζητάμε για τα clusters και καλό θα ήτανε να υπάρχουν ε, ομάδες εργασίας σε κλάστερς που να επεξεργάζονται τα θέματα αυτά. Επίσης όσον αφορά την τροπολογία 22. Ήθελα ε, να δημοσιευθεί μία μορφή που να είναι πιο φιλική ε, για τον αναγνώστη διότι εδώ ζητάτε ε, ένα δελτίο τύπου συγχρόνως με τον πίνακα βαθμολόγησης. Νομίζω λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να παρουσιάσει μία ανακοίνωση τύπου πιο φιλική για τον αναγνώση ε, για να μπορέσει να εφαρμόσει την ε, οδηγία. Και αυτή είναι η δεύτερη πρότασή μου. Και βέβαια ο στόχος μου είναι να επιστήσω την προσοχή σε αυτό το πίνακα βαθμολόγησης και να αυξήσουμε και την πίεση. Διότι ο πίνακας βαθμολόγησης είναι ένας θαυμάσιος τρόπος για να ε, εφαρμοστούν ε, οι μέθοδοι συχνά. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κυκλοφορεί με, έχοντας ε, στην τσάντα της αυτούς τους πίνακες βαθμολόγησης και θα ήθελα να ευχαριστήσω και την κυρία Τούν για την εξαιρετική συνεργασία. Ωραία. Ο κύριος Τριανταφυλλίδης δεν παρίσταται. Περνάμε λοιπόν στους υπόλοιπους που έχουν ζητήσει το λόγο. Η κυρία Γκέπχαρτ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Εισηγήτρη για την καλή δουλειά και τη και το σκιώδη εισηγητή μας, διότι από ό,τι έχω παρακολουθήσει η συνεργασία ήταν πολύ θετική και πολύ καλή, οπότε κοιτώ σχετικά με την ε, τροπολογία 1, διότι με τη γενική μετάφραση εγώ δεν συμφωνώ, ούτε η Λίντα θα συμφωνήσει, υπάρχει κάποιο λάθος στη μετάφραση νομίζω, και πρέπει να φροντίσουμε να διορθωθεί τουλάχιστον η μετάφραση. Δηλαδή το γαλλικό κείμενο είναι το ισχύον για την ψηφοφορία και πρέπει να είναι σαφές ε, περί την ομιλούμε. Διότι δεν λέμε ότι πρέπει να αγοράζει κανείς τις φθηνότερες υπηρεσίες αλλά πρέπει να είναι και πολύ ψηλή ποιότητα και όσο το δυνατόν πιο συμφέρουσε. Κάπω έτσι θα έπρεπε να μεταφραστεί και όχι όπω αναφέρεται εδώ. Και αυτό είναι σαφές. Ζήτησα όμως το λόγο, λόγω της τροπολογίας 19 την οποία δεν μπορεί να υπερψηφίσει η πολιτική μας ομάδα και το είπε και η κυρία Ρούιλε διότι εις ε, της Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Ενώσεως δεν αναφερόμαστε μόνο στον ανταγωνισμό σε υγιή και δίκαιο ανταγωνισμό αλλά με την είσοδο σήμερα ε, σε ισχύ της ε, Συνθήκης Λισαβόνας βλέπουμε ότι υπάρχουν και άλλα βασικά συστατικά στοιχεία και γι' αυτό πρέπει να συμφωνήσουμε για μια εσωτερική αγορά ενώ τα άλλα θέματα τα οποία μπορεί να είναι πολύ σημαντικά για τον πολίτη δεν, δεν περιλαμβάνονται σε αυτό το κείμενο και γι' αυτό δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Γι' αυτό και δεν το είχαμε υπερψηφίσει στην προηγούμενη θητεία και μεταξύ δεν αλλάξαμε την άποψή μας. Πρέπει να πω για την πολιτική μου ομάδα, διότι το συζητήσαμε και σήμερα το μεσημέρι, αυτή η τροπολογία. Εάν υπερψηφιστεί, εμείς δεν θα ε, ψηφίσουμε και δεν θα δεχθούμε ολόκληρο το κείμενο διότι δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι ε, δεν θα είναι στο επίκεντρο ο πολίτης και θα είναι οι επιχειρήσεις και αυτό λέγεται εδώ είναι λοιπόν κάτι το οποίο δεν μπορούμε να δεχτούμε. Ευχαριστώ. Δίνω το λόγο τώρα στον κύριο Πουπάκη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Ντόν για την πολύ καλή δουλειά της να την ευχαριστήσω για τη συνεργασία της και που έκανε δεχτές τις τροπολογίες μου. Πράγματι, ο πίνακας αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς είναι πολύ σημαντικός, καθώς συμβάλλει στη δημιουργία μιας πιο αποτελεσματικής εσωτερικής αγοράς. Μέσα από τις τροπολογίες που υποστήριξα, κυρίως μεγαλύτερη συνεργασία και συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων και των άλλων φορέων, μεταξύ των οποίων και των κοινωνικών εταίρων, στους οποίους θεωρώ πολύ σημαντικού καθώς μέσα από τα δίκτυα πληροφόρησης που διαθέτουν μπορεί να γίνουν ένας ακόμα διάβλος πληροφόρησης των καταναλωτών. Επιπλέον υποστήριξα ότι τα κράτα-μέλη πρέπει να αξιοποιήσουν τις υφιστάμενες κατευθυντήριες γραμμές για το μέσο ανταλλαγής των βέλτιστων πρακτικών, όπως και τη σημασία του ανοιχτού διαλόγου, καθώς και μια πιο στενή συνεργασία στο Εθνικό Κοινοβούλιο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με σκοπό να αντιμετωπιστεί άμεσα και με ακρίβεια το υφιστάμενο έλλειμμα μεταφοράς νομοθεσίας. Τέλος, πιστεύω ότι οι εμπειρίες από το Solvit πρέπει να ενσωματώνονται στην εθνική χάραξη πολιτικής καθώς και στη χάραξη της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πάλι να ευχαριστήσω την κυρία Τον. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Wang. Θέλω απλά να προτείνω μια προφορική τροπολογία. Δεδομένης αντίδρασης συναδέλφου. Όντως, ακόμα και αν δεν είναι η καλύτερη τη μετάφραση, να μην υπάρχει καμία αμφισημία, προτείνω να αφαιρέσουμε το τελευταίο όρο της προβληματικής φράσης, δηλαδή θα πρέπει να λέει οι καταναλωτές μπορούν να προμηθευτούν ε, ποιοτικά αγαθά και υπηρεσίες και εκεί αφαιρούμε το au moindre prix, δηλαδή στη χαμηλότερη δυνατή τιμή. Πράγμα που είναι σωστό. Ε, εξάλλου δεν είμαι και ένθερμος υποστηρικτής ε, του low cost, του χαμηλότερου δυνατού κόστους. Αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι η ποιότητα. Ωραία. Περνάμε τώρα στην Κομισιόν και την κυρία Μόρκ. Είναι ο κύριος Μόρκ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η Κομισιόν, όπω είπε και παλιότερα καλωσορίζει την έκθεση τη κυρία Τούν και η συνεργασία που είχαμε μαζί τη ήταν υποδειγματική. Όσον αφορά τις τροπολογίες, επίση τις καλωσορίζουμε. Έχουμε κάποιες μικρές ε, ανησυχίες. Αν επιτρέπετε θα τις αναφέρω εν συντομία. Η πρώτη αφορά την ε, τροπολογία 2 που λέει δημοσίευση του πίνακα βαθμολογίας, μπορεί, πίνακα αποτελεσμάτων στις τοκές αγορά μπορεί να συνεισφέρει, ενώ κατά την άποψή μας συνεισφέρει. Και είναι πολύ σημαντικό να στείλουμε αυτό το μήνυμα ξεκάθαρα, ότι δηλαδή η πίεση μεταξύ άμυλα ανάμεσα στους ε, ε, στα κράτη-μέλη ε, θα δώσει κάποια αποτελέσματα. Θέλουμε λοιπόν να λέει συνεισφέρει και όχι μπορεί να συνεισφέρει. Στην ε, τροπολογία 17 λέει πως ε, ο πίνακας αποτελεσμάτων θα πρέπει να δημοσιεύεται με την ίδια συχνότητα. Αυτό δεν είμαστε κατά βέβαια. Αυτή τη στιγμή ο πίνακα αποτελεσμάτων τη εσωτερική αγορά ε, ε, δημοσιεύεται δύο φορέ το χρόνο, ενώ ο πίνακα αποτελεσμάτων για του καταναλωτέ μία φορά. Όμω θα θέλαμε να διατηρήσουμε τη δύο φορέ το χρόνο τον πίνακα αποτελεσμάτων τη εσωτερική αγορά ε, και δεν είναι δύσκολο για μα να διπλασιάσουμε και τη συχνότητα έκδοση δημοσίευση των αποτελεσμάτων για του καταναλωτέ. Για την 21. Σε κάποιο βαθμό υπάρχει επικάλυψη για το τι δημοσιεύεται στην ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας και την ε, πίνακα αποτελεσμάτων. Τονίζουμε την ετήσια έκθεση, όμως εδώ καλύπτεται όχι μόνο η εσωτερική αγορά, αλλά μια ολόκληρη, ένα ολόκληρο φάσμα δραστηριοτήτων της Επιτροπής Είναι, και μπαίνει σε πολύ περισσότερες λεπτομέρειες με διάφορα θέματα τα οποία δεν ε, αφορούν απαραίτητο στα θέματα που καλύπτει ο πίνακα αποτελεσμάτων τη εσωτερική αγορά. Φαίνεται δηλαδή εδώ ότι υπάρχει επικάλυψη, ενώ δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο στην πραγματικότητα. Με την τροπολογία 22. Να σας πω ότι ναι, εκδίδεται ε, ε, συνέντευξη τύπου κάθε φορά που εκδίδεται και ο πίνακας αποτελεσμάτων. Προσπαθούμε να το κάνουμε όσο γίνεται πιο ευανάγνωστο. Αυτό που είναι σημαντικό για να υπάρξει μεγαλύτερη διάδοση των πινάκων αποτελεσμάτων είναι οι γλωσσικές εκδοχές και αυτό θα το δούμε τον επόμενο χρόνο. Μήπως μπορούμε να το δημοσιεύσουμε και σε άλλες γλώσσες και όχι μόνο στα αγγλικά. Και το ανακοινωθέν τύπου το κάνουμε κάθε φορά. Για την τροπολογία 26. Νομίζω πως θα ήταν καλή ιδέα, αν, το αν συμφωνεί το Κοινοβούλιο, να αναφερθούμε στο συστάσεις του 2004 για την μεταφορά, που συμπεριλαμβάνει ένα κατάλογο καλύτερων πρακτικών στον τομέα της μεταφοράς νομοθεσίας. Και αυτό που είναι σημαντικό είναι όχι τόσο μόνο να τονίσουμε τις ε, καλές πρακτικές, αλλά να δούμε αν αυτές εφαρμόζονται στα κράτη-μέλη. Και έχουμε χρησιμοποιήσει τον πίνακα των αποτελεσμάτων για το μετρήσουμε αυτό στο παρελθόν και μπορούμε και να το ξανακάνουμε στο μέλλον. Και μετά για την τροπολογία 33 θα ήθελα να πω τα εξής. Τα εργαλεία που προβλέπονται από την οδηγία για τις υπηρεσίες και ιδιαίτερα τα σημεία επαφής έχουν πολύ διαφορετικούς ρόλους να παίξουν και κατά συνέπεια διάφορα είδη πληροφόρηση θα πρέπει να δίνονται στις επιχειρήσεις κάθε φορά. Είναι σαφές ότι τόσο η ότι και τα δύο αυτά γραφεία είναι, έχουν στόχο να δίνουν πληροφορίες Δεν επικαλύπτονται αυτοί οι δύο μηχανισμοί, ωστόσο, είναι συμπληρωματικοί και γι' αυτό η τροπολογία 33 μπορεί να είναι λίγο παραπλανητική από αυτού. Τέλος, θα ήθελα να πω για την τροπολογία 36, για το Solvit και την έκκληση να γίνουν περαιτέρω προσπάθειες για να γίνει πιο ορατό το Solvit στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τους πολίτες. Συμφωνούμε εδώ και ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις, γιατί αν δούμε το Solvit το 2009, είναι σαφέ πω οι πολίτε το έχουν χρησιμοποιήσει πολύ, ενώ οι επιχειρήσεις όχι όσο θα θέλαμε. Άρα υπάρχει μια πρόκληση όσον αφορά την ορατότητα. Το θέμα είναι α, πού ακριβώς έγκυται η πρόκληση. Είναι θέμα της Κομισιόν ή των κρατών. Κατά την άποψή μας είναι περισσότερο θέμα των κρατών μελών. Αυτοί που ακριβώ κράτη-μέλη. Κατά την άποψή μας λοιπόν αυτή είναι η προκληση ειναι θεμα τη κομισιον η των κρατων κατα την αποψη μα ειναι περισσοτερο θεμα των κρατων μελων αυτοι που πρόκληση. Θα ήταν χρήσιμο λοιπόν να αντικατοπτρίζετε καλύτερα η πραγματικότητα στην τροπολογία αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Να δώσω το λόγο στην κυρία Γκέπχαρτ. Ε, αισθάνθηκα ότι με προκάλεσαν τα τελευταία σχόλια του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρέπει λοιπόν να σας πω ότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να δεχτώ. Όντως είναι κάτι το οποίο πρέπει να προσφερθεί από τα κράτη-μέλη και είναι μια παροχή υπηρεσιών των κρατών μελών η οποία έτσι έχει προβλεφθεί. Πρέπει όμως η τροπολογία αυτή να υπερψηφιστεί, διότι στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως έχουμε εξαιρετικά μία έκτακτη γραμμή για να μπορεί να έχει κονδύλια Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διαφημίζει, να οργανώσει δηλαδή μία εκστρατεία ενημέρωση στα κράτη-μέλη. Και εγώ δεν τη βλέπω. Και διαβάζω όταν ε, συζητάμε για τον προϋπολογισμό και όταν ε, κάνουμε την, ε, τον έλεγχο για το 2008 ότι ελάχιστα κονδύλια έχουν διατεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θεωρώ είναι ντροπή, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αντίθετη σε αυτή τη γραμμή του προπολογισμού και νομίζω ότι δεν υπάρχει πολιτική θέληση να εφαρμόσουμε αυτά τα οποία έχει απαιτήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γι' αυτό και υπάρχει αυτή η τροπολογία και είναι σημαντική σε αυτά τα συμφραζόμενα. Ωραία, δίνω το Σας ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Τούν. Τροπολογία 1 χαμηλότερη τιμή. Υπήρξε μια προφορική τροπολογία, δεν το κατάλαβα. Lower price είπε. Ναι. Πρέπει να λάβουμε υπόψη την πρόταση του συναδέλφου Hang Νομίζω ότι είναι μια λύση για τη συζήτησή μας, αν εξεφράσουμε το δεύτερο κομμάτι της πρότασης που λέει να αγοράζουν αγαθά και και να δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας. Τι λένε οι φιλελεύθεροι γι' αυτό. Αυτό πρότεινε στην προφορική του τροπολογία. Να ξεφορτωθούμε το δεύτερο κομμάτι. Ναι. Όχι, έχουμε διαφορετική θέση, κυρία Γκέπχαρτ. Έχουμε προτείνει ε, μόνο στα γερμανικά να διαγραφούν τρεις λέξεις, όχι μία παράγραφος, το, οι λέξεις υπερβολικά χαμηλές τιμές. Μόνο αυτές οι τρεις λέξεις ζητάμε να διαγραφούν. Οπότε αυτή είναι η προφορική τροπολογία. Εντάξει. ακούγοντας και την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση επί του θέματος, Έχουμε και την τροπολογία 19, αλλά ο Μάλκον δεν είναι εδώ, άρα θα επανέλθουμε. Επιμένει σε αυτήν την τροπολογία του. Από ό,τι γνωρίζω, το Κοινοβούλιο έχει ήδη προτείνει, είχε κάνει την ίδια πρόταση και την προηγούμενη φορά. Νομίζω λοιπόν ότι η εσωτερική αγορά και η αξιολόγηση της είναι πολύ σημαντική για την περαιτέρω εξέλιξη, γι' αυτό και θα ήθελα να την διατηρήσω. Τώρα, η τροπολογία 26 συζητήθηκε. Εάν δηλαδή ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, ε, εντοπίσει τις βέλτιστες πρακτικές υπό τη υπογραπτή μορφή ή υπό τις καλύτερες συνθήκες. Πάντοτε μπορούμε να το αναλύσουμε πιο βαθιά και δεν υπάρχει επαρκή στάφτιση. Νομίζω όμως ότι είναι παρανόηση. Πού είναι ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όταν λοιπόν ζητάτε από τα κράτη-μέλη και λέτε ότι δεν είναι ευθύνη του, της Επιτροπής αλλά των κρατών μελών, Γι' αυτό έχω προτείνει και αυτό το φόρουμ της εσωτερικής αγοράς. Είναι ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υποκινήσει τα κράτη-μέλη, να συντονίσει την εργασία, να προσφέρει περισσότερες πληροφορίες, να οργανώνει συζητήσεις και η τροπολογία 33 αναφέρεται στην σαφέστατη απαρίθμηση όλων των πληροφοριών και των ιστοσελίδων που έχουμε. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο νομίζω μπορεί να βελτιώσει την δράση ενημέρωσης. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε πιο ο διαφανείς ε, πληροφορίες ασχέτως των μεθόδων. Πρέπει να γίνει πολλή δουλειά και γι' αυτό εγώ θα ήθελα να αφήσω την τροπολογία αυτή ως έχει, όπως ε, ισχύει και για την ε, τελευταία τροπολογία. Αντιλαμβάνουμε ότι αν αποσύρουμε τις τρεις λέξεις σαν προφορική τροπολογία στην αρχή, δεν θα έχουμε συμφωνήσει όσο το όσο, όσον αναφορά τα υπόλοιπα και μπορούμε να προχωρήσουμε εις ε, την ε, ε, στην Μάλιστα, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω ότι στην Κομισιόν αν θέλει να παρέμβει και πάλι για αυτό το θέμα ή αν, αν δεν το θεωρείτε σκόπιμο μπορούμε να συνεχίσουμε. Ε, ίσως εν συντομία να πούμε τα εξής. Δεν είναι ένα θέμα ε, για να αποφύγει η Επιτροπή την ευθύνη της επίλυσης. Ίσως ε, θα μπορεί να γίνει μια αναφορά τόσο στην Επιτροπή όσο και τις χώρες. Ε, το Solvit είναι μια ξεκάθαρη προτεραιότητα για την Επιτροπή. Πρόκειται για ένα άλλο θέμα. Η τοπικές αρχές είναι πιο κοντά και οι περιφερειακές αρχές πιο κοντά στον πολίτη και γνωρίζουν καλύτερα, να, μπορούν καλύτερα να φτάσουν τις ανάγκες των πολιτών. Η Επιτροπή δεσμεύεται στην πρόθεση των δραστηριοτήτων. Αλλά αν θέλετε να υπάρχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα ε, στο δινεκές, ε, νομίζω ότι είναι αναγκαίο να καλέσουμε τις χώρες ε, μέλη να δεσμευθούν εδώ, να αναλάβουν ίδιες κάποια δράση. Μάλιστα, δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις. Ναι, παρακαλώ. Νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε να εισήσουν και τα δύο. Δηλαδή οι επιτροπές και οι χώρες μέλη, να το διατυπώσουμε έτσι, νομίζω ότι αυτό μας βρίσκει σύμφωνος. Η κυρία Τούν. Ναι, θα ήθελα να καλέσω την Επιτροπή ε, να, όχι να αισθανθεί ότι είναι μια μορφή προς την εξαιρετική εργασία που έχει επιτελέσει. Είναι μάλλον μια ε, πράξη έγκριση, αναγνώριση τα όσα κάνατε και έχουμε το δυναμικό μιας περαιτέρω ε, εργασίας. Αλλά βεβαίως και οι χώρες μέλη θα πρέπει να συμμετάσχουν και καλούμε τους ε, συναδέλφους ε, από τις χώρες μέλη να συμμετάσχουν στο θέμα αυτό. Και πραγματικά θα συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε το θέμα αυτό και τις προσπάθειές μας. Αν δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις, να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και τους Κεώδης για την εξαιρετική τους ε, εργασία και για την ανταλλαγή αυτή απόψεων που ήταν πολύ χρήσιμη. Να θυμίσω πως αύριο θα ψηφίσουμε το πρωί στις 10 και θα έχουμε ψηφοφορία στην Ολομέλεια την 1η Μαρτίου μαζί με τις εκθέσεις για το Solvit και για το πλαίσιο αξιολόγησης των ε, αγορών αγαθών καταναλωτικών. Ωραία, λοιπόν, μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Ασφάλεια ανεφοδιασμού σε φυσικό αέριο. Η κυρία Καρνιέτε έχει το λόγο. Thank you, Madam Chairwoman. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι πραγματικά λυπούμε που δεν έχω δυνατότητα να μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα, γιατί είναι μια ωραία γλώσσα, δεν είναι μόνο τα αγγλικά και άλλες γλώσσες ωραίες. Αλλά θα ξεκινήσω αυτό που έχω στη διάθεσή μου. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι το σχέδιο κανονισμού έτσι όπως έχει παρουσιαστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν πραγματικά εξαίρετο και ήταν χαρά μας να συνεργαστούμε με τις ε, υπηρεσίες της Επιτροπής. Κατά δεύτερο λόγο θα ήθελα να πω ότι είμαι πολύ ευτυχής που πετύχαμε μια πλατιά συνένεση μεταξύ των πολιτικών ομάδων ε, σε όλες τις συμβαστικές, ως προς που υποστηρίζονται από το ΕΛΚ, από το ΑΛΔΕ, του Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Δύο συμβαστικές τροπολογίες, ε, για δύο συμβαστικές έχουμε και το ECR και το ΓΚΟΕ. E. Επίσης, ε, θα ήθελα να πω ότι ήταν μια εξαιρετική συνεργασία με τις χώρες ε, μέλη στην Επιτροπή ΙΜΚΟ από όλες τις πολιτικές ομάδες και θα ήθελα επίσης να επεκτείνω τις ευχαριστίες μου και προς τη Γραμματεία ε, ήταν μια χαρά να ε, συνεργαστούμε μαζί τους. Ε, τώρα, ποιες είναι οι βασικές συμφωνίες. Καταρχήν, θα ήθελα να πω ότι επεξεργαστήκαμε μια, έναν επαρκή ορισμό των πελατών. Υπάρχει μια ξεκάθαρη διάκριση μεταξύ ευάλωτων πελατών και να και στις χώρες μέλη να αποφασίσουν ποιοι είναι και να παράσουν κάποιες εγγύσει για αυτή την ομάδα. Επίσης, συμπεριλαμβάνεται μία αναφορά στην ελεγγύη. Και αυτό είναι ιδιαίτερο σημαντικό υπό το πρίσμα της ε, έναρξης ισχύω της συνθήκη της Λισαβόνας. Ο κανονισμός τώρα θα πρέπει να βασίζεται στο άρθρο 194, το οποίο λέει ότι η ενέργεια θα πρέπει να τεθεί στην υπηρεσία του πνεύματος αλληλεγγύης. Ε, όλα είναι βεβαίως εργαλεία που βασίζονται στην αγορά, ακόμα και σε περιόδους κρίσης. Επίσης τονίζουμε την ευθύνη των εθνικών εταιριών εφοδιασμού με φυσικό αέριο, ε, ιδιαίτερα σε ε, περιόδους έκτακτης ανάγκης. Οι τροπολογίες αυτές αντανακλούν επίσης τη σημασία των υποχρεώσεων του δημόσιου τομέα. Κάνουν μια διάκριση μεταξύ των προστατευόμενων ε, καταναλωτών και των ε, ευάλωτων καταναλωτών. Και επίσης είχαμε τη δυνατότητα να ορίσουμε μια κοινή θέση σε σχέση με την ε, πρόληψη μιας υπερβολικής ε, τιμολόγησης. Τώρα, μιλώντας για τροπολογία υπαρθμών 1, η τροπολογία αυτή ορίζει το, την εμβέλεια των προστατευμένων καταναλωτών, περιλαμβάνουν τα νοικοκυριά, τα σχολεία κλπ. Επίσης, το εναρμονισμένο φάσμα των προστατευμένων καταναλωτών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπενθυμίζει για τους ευάλωτους καταναλωτές ότι θα πρέπει η ομάδα αυτή να ορίζεται από την κάθε χώρα μέλος ξεχωριστά. Αυτή η διάκριση μεταξύ προστατευμένων και ευάλωτων καταναλωτών ε, διέπει, ε, διαπερνά ολόκληρο το κείμενο του κανονισμού ε, και η ομάδα των προστατευμένων καταναλωτών περιλαμβάνει και τους ευάλωτους καταναλωτές. αφορά επίσης την αξία της, των πρώτων υλών, ε, τονίζει τη σημασία πρόληψης της υπερβολικής ε, αύξησης των τιμών, ενώ η Συμβαστική Τροπολογία Υπαριθμών 3 λέει ότι είναι η ευθύνη των χωρών μελών να ενημερώσουν του καταναλωτέ για το δικαίωμα που έχουν να προστατεύονται κατά τι περιόδου κρίση και προσθέτει ότι η αύξηση του κόστους για τις ευάλωτες ομάδες στις περιόδους ε, κρίσης. Ε, θα πρέπει να αντισταθμίσετε. Τέλος, η συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 4 επιτρέπει στις χώρες μέλη να ζητούν ε, έκτακτη παρέμβαση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφαρμόζοντας μια διαδικασία εκπαλήθευσης εκ μέρους της Επιτροπής. Τώρα, ποιες είναι οι βασικές αρχές για όλες αυτές τις τροπολογίες όσον Καταρχήν, εναρμονίζονται τα στάνταρτς ε, εφοδιασμού σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τονίζει το ρόλο των ε, μηχανισμών της Ένωσης για την πρόληψη των κρίσεων και ε, η παρέμβαση στην αγορά θα πρέπει να αξιοποιείται μόνο εφόσον έχουν εξαντληθεί όλα τα άλλα μέσα. Ε, ενισχύει την αρχή της ελεγγύης προς ευάλωτους ε, καταναλωτές και ενισχύει την ανάγκη ελεγγύης μεταξύ των χωρών μελών. Και εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Τεσκόφσκι για τη δική του εισφορά, υπενθυμίζοντας ότι η συνθήκη της Λισαβόνας έχει τεθεί σε ισχύ και ο κανονισμός θα πρέπει να βασίζεται στο άρθρο 194 της συνθήκης. Και αυτό το οποίο είναι σημαντικό για τον καθένα από εμά είναι να έχει μια έγκαιρη ενημέρωση. Ο ρόλος της Επιτροπής στην παρακολούθηση της συμμόρφωσης ε, των ε, συμφωνιών για τον αναθωρισμό με φυσικό αέριο έχει τεθεί σε ισχύ. Επίσης, θέλω να σε επενθυμίσω ότι πολλές τροπολογίες δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Επιτροπής ΣΥΜΚΟ και θα ήταν καλύτερο να κατατεθούν και να συζητηθούν στην στην Επιτροπή Ήτρε. Γι' αυτό ε, αναμένω τη συνέχεια αυτής της συζήτησης με την Ήτρε. Και λοιπόν θα πρέπει να πω ότι ορισμένε τροπολογίες δεν συμφωνούν απολύτως με το πνεύμα του κανονισμού. Για παράδειγμα έπρεπε να απορρίψουμε ορισμένε από αυτές. Και τώρα ποια είναι τα επόμενα βήματα. για τη δική μας Επιτροπή έχουμε την αυριανή ψηφοφορία. Η εργασία μας έχει σχεδόν περατωθεί και θα ήθελα πραγματικά να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Σβάμπ, τους κοιόδες μου εισηγητές, τον κύριο Σίγκετς, τον κύριο Μάντες και τον κύριο Τρενταφυλλίδη. Και ιδιαιτέρως από την ε, ΙΜΚΟ, ε, τον κύριο Βαντελα από το προσωπικό της ΙΜΚΟ. Ε, σας ευχαριστώ πολύ. σας ευχαριστώ για την πολύ εμπεριστατωμένη σας έκθεση. Να δώσουμε το λόγο στον σκιώδη συγγετή, τον κύριο Σίβιτς. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Αύριο θα ψηφίσουμε. Θα ψηφίσουμε τις τροπολογίες αυτές μετά από μια μακρά και έντονη συζήτηση θα ήθελα να πω με, προς μεγάλη μου κανοποίηση ότι παρά το γεγονός ότι ξεκινήσαμε την εργασία αυτή με διαφορετικές προπτικές, τελικά καταλήξαμε σε μια αρκετά ακριβή διατύπωση των απόψεών μας και τον ορισμό της προστασίας των καταναλωτικών αγαθών. Σε συγκεκριμένη περίπτωση, όταν μιλάμε για την παροχή ενέργειας, και την παροχή φυσικού αερίου αγγίζουμε ένα πολύ περίπλοκο θέμα. Έχει ήδη αναφερθεί στην αίθουσα αυτή επανειλημμένος και διάφορες άλλες επιτροπές έχουν γνωμοδοτήσει επί του θέματος αυτού. Έχω την εντύπωση ότι αν κανείς ρωτήσει Τι σημαίνει ακριβώς ασφάλεια ανεφοδιασμού σε φυσικό αέριο όσον αφορά την προστασία των ε, καταναλωτικών αγαθών θα μπορούσε κανείς να ακολουθήσει διάφορες προοπτικές. Από τη μια πλευρά ο τελικός καταναλωτής πρέπει να είναι βέβαιος ότι θα έχει φυσικό αέριο και από την άλλη πλευρά δεν μπορεί κανείς να τον εξαπατήσει όσον αφορά την τιμή και γενικά τον τρόπο παροχής του φυσικού αερίου. Άλλοι, λοιπόν οι προτεραιότητες που είχαμε θέσει έχουν επιτευχθεί, ειδικά οι διατάξεις που εγγυώνται και ορίζουν τους προνομιούχους ή προστατευόμενους χρήστες. Μιλάμε για αυτούς που προστατεύονται στον υψηλότερο βαθμό και που πραγματικά δεν, αν, δεν αποδυναμώνουμε την έννοια του καταναλωτή που πρέπει να προστατευτεί. Πριν από την κρίση ε, είχαμε πρόβλημα με τις τιμές του φυσικού αερίου ε, και η ομάδα μου θα υποστηρίξει τις πέντε συμβιβαστικές τροπολογίες. Να σχολιάσω και το εξή. Πέρα από τι βασικέ τροπολογίε, έχουμε επίση υποβάλει κάποιε ίσονε σημασίε που δεν είναι τόσο αντιφατικέ, αλλά όταν μιλάμε για ενεργειακή πολιτική, πολιτική που σχετίζεται με το συγκεκριμένο ψήφισμα, είναι καλύτερο να κατανοήσουμε τη λέξη αλληλεγγύη ως αμοιβαία ευθύνη, αμοιβαία παροχή υπηρεσιών, μεταξύ μας και μπορούμε ειλικρινά να πούμε ότι στο τομέα της συνεργασίας ε, στην ενέργεια η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε ένα νηπιακό στάδιο. Τώρα μόλις αρχίζουμε να μιλάμε για το πώς μπορούμε να προστατεύσουμε οι μεν τους δε σε περίπτωση απειλής. Ελπίζω πως ε, η Επιτροπή μας, που είναι υπεύθυνη για την εσωτερική αγορά και για την προστασία του καταναλωτή, θα ξανασχοληθεί με τα θέματα αυτά και πιστεύω πως κάναμε πολύ καλή δουλειά αυτή τη φορά. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια, αλλά και τους ε, συναδέλφους ε, σκεώδης εισηγητές από άλλες ομάδες, αλλά να ευχαριστήσω και την γραμματεία μας, η οποία εκπλήρωσε το βαρύ καθήκον να συνδυάσει τις σκέψεις ανθρώπων που δεν ε, ταυτίζονται πάντοτε. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Μάντερς που είναι σκιώδης συζητής. Thank you very much, Chair. Um, I don't want, well, of course, uh, I, want to thank uh, Mr. Calniete for the, uh, for the, to cooperate with. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια γιατί έδειξε μεγάλο πνεύμα συνεργασίας για την ε, εξέταση των τροπολογιών. Υποβάλαμε νέα τροπολογίες και υπήρξε και μια παρεξήγηση για το κατά πόσο τούτη η Επιτροπή ήταν αρμόδια ή όχι, αν έπρεπε να γνωμοδοτήσει ή όχι. Ακόμα συζητείτε το θέμα και ψηφίζουμε γι' αυτό αύριο. Οι δικέ μα τροπολογίε αφορούν την εσωτερική αγορά και του καταναλωτέ. Για παράδειγμα, όταν μιλάμε για την ε, μεταγραφή της οδηγίας για το φυσικό αέριο, εγώ νομίζω πως είναι προς το συμφέρον των καταναλωτών και είναι σημαντικό για τους καταναλωτές. Όταν μιλάμε για την ε, σύνδεση του Ευρωπαίου νομοθέτη, είναι και αυτό υπέρ της βελτίωσης της εσωτερικής αγοράς. Αν τα δίκτυα δεν είναι συνδεδεμένα, τότε δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ε, αλληλεγγύη για τους άλλους καταναλωτές, γιατί δεν υπάρχει δίκτυο από τη μια χώρα στην άλλη. Νομίζω λοιπόν πως ε, όλα αυτά είναι τμήμα της εσωτερικής αγοράς και είναι και προς το συμφέρον του καταναλωτή. Ελπίζω ότι θα μπορέσετε να υποστηρίξετε τις 9, 13, 14, 43 και 63 τροπολογίες. Οι αιτιολογήσει τους ε, έχουν ε, εξαφανιστεί, δεν ξέρω γιατί, ίσως θα μπορούσαμε να τις προσθέσουμε για αύριο, γιατί αυτό δίνει μια καλύτερη κατανόηση όταν ε, εξηγούμε γιατί είναι σημαντικές οι τροπολογίες αυτές. Είναι σημαντικό να δούμε ότι όταν η εσωτερική αγορά λειτουργεί ομαλά είναι προς το συμφέρον των καταναλωτών. Και όταν μιλάμε για αλληλεγγύη χρειάζεται πάνω κάτω ένα ολοκληρωμένο δίκτυο σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και το λέμε αυτό για την οδηγία του φυσικού αερίου, αλλά αν τα κατημέλη δεν μεταφέρουν αυτήν την νομοθεσία στην εθνική τους νομοθεσία, έχουμε δυσκολίες. Γι' αυτό και σκεφτόμουν πώς θα μπορέσουμε να επιβάλλουμε στα κρατη να εφαρμόσουν ή να μεταφέρουν την οδηγία για το φυσικό αέριο έτσι ώστε όταν θα εφαρμοστεί αυτή η οδηγία να εφαρμοστεί και η οδηγία για το φυσικό αέριο ταυτόχρονα. Για την ώρα δεν γίνεται μεγάλη προσπάθεια για την ε, χρήση της οδηγίας. Τέλος, μπορώ να υποστηρίξω τις συμβαστικές τροπολογίες που συνέταξε η κυρία Καλνιέτη, η γήτρια, και αυτές τις υποστηρίζουμε λοιπόν και σας ευχαριστώ που κάνατε συμβαστικές τροπολογίες. Ελπίζω και αυτό είναι σημαντικό ότι θα μπορέσουμε να δώσουμε ένα μήνυμα στην αρμόδια από τις επιτροπή γιατί Συνήθω ε, δεν λαμβάνουν πολύ υπόψη του νομοδοτήσεις των άλλων επιτροπών και τι συμβουλέ του. Ελπίζω πω θα μπορέσουμε να του πείσουμε πω μιλάμε όντω για την εσωτερική αγορά και την προστασία των καταναλωτών, αν μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό. Η, η συγγήτριά μας δηλαδή, αν μπορέσει να τα καταφέρει και να πείσει του συναδέλφου στην Επιτροπή Ήτρε, θα είναι πολύ θετικό. Αυτά ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ κύριε Μάντερς και τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Βούλεν. Δεν ήμουν ε, ε, σκιώδης, αλλά δεν είναι εδώ σκιώδης και γι' αυτό δεν θα λάβω το λόγο, διότι ήδη έχουμε ξεπεράσει την ώρα. Δεν θέλετε δηλαδή να παρέμβετε, εντάξει. Ωραία, λοιπόν, να δώσω το λόγο στον κύριο Τριανταφυλλίδη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την προθυμία της να συζητήσει μαζί μας ε, το όλο ζήτημα και να συνεργαστούμε σε ένα πολύ καλό και θετικό κλίμα. Η δική μας η ομάδα έχει καταθέσει μια σειρά τροπολογιών. Μερικές από αυτές έχουν ληφθεί υπόψη στην ε, καταρτισμό των ε, compromise amendments και θα προσυπογράψουμε μερικές από αυτές τις compromise amendments αλλά έχουμε και άλλες ε, τροπολογίες που έχουμε υποβάλει ε, και όλες αυτές βασίζονται πάνω σε δύο βασικές σκέψεις. Πρώτον, θέλουμε να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη-μέλη να συμπεριλάβουν στους προστατευόμενους πελάτες ομάδες της οικονομίας, τις οποίες αυτά τα κράτη-μέλη δηλαδή θεωρούν ως τις πιο ευάλωτες. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να διατηρήσουν τον ενεργό τους ρόλο στην λήψη αποφάσεων και να διασφαλίσουν την ασφάλεια εφοδιασμού κατά τον εφοδιασμό της αγοράς με φυσικό αέριο. Και η δεύτερη μας σκέψη αφορά στα μέτρα που λαμβάνονται σε περιόδους έκτακτης ανάγκης. Πιστεύουμε ότι τα μέτρα αυτά θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να ανταποκρίνονται στην τρέχουσα κρίση. Βασικό κριτήριο δεν μπορεί να είναι ο βαθμός ανταπόκρισης στην εσωτερική αγορά, αλλά η αποτελεσματικότητα στη στήριξη των καταναλωτών. Ως εκ τούτου, μερικές από τις τροπολογίες μας που έχουμε καταθέσει καθορίζουν ότι η αρμόδια αρχή πρέπει να εννοείται πάντα η αρμόδια εθνική ρυθμιστική αρχή. Γιατί οποιαδήποτε παρέκκληση αυτού του κανόνα στρεβλώνει την ουσιώδη λειτουργία και σκοπό ύπαρξη τη αρχή ω ανεξάρτητου φορέα που μεριμνά για το συμφέρον των καταναλωτών. Επιπλέον έχουμε καταθέσει άλλε τροπολογίε που αφορούν το δικαίωμα του κάθε κράτου να εξασφαλίσει τα οικονομικά του συμφέροντα το οποίο δικαίωμα δεν μπορεί να τίθεται υπό την κυδαιμονία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η σύναψη διακυβερνητικών συμφωνιών πιστεύουμε είναι κρατικό ζήτημα και εγκρίνεται μόνο από εθνικά κοινοβούλια και γι' αυτό τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν τον πρωταρχικό ρόλο στη σύναψη διακρατικών συμφωνιών. Και τέλος, αγαπητοί συνάδελφοι, οι άλλες προπολογίες που έχουμε καταθέσει έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν ότι τα μέτρα για αντιμετώπιση των συνθήκων έκτακτη ανάγκη δεν θα επάγονται αποκλειστικά στου κανόνε τη αγορά και των συμφέρων των επιχειρήσεων, αλλά κύρια στι ανάγκε των καταναλωτών. Αυτά και ευχαριστώ πολύ. ευχαριστώ πολύ. Θέλει κάποιος άλλος να πάρει το λόγο. Αλλιώς θα δώσω το λόγο στην Κομισιόν. Στον κύριο Μπενουά. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν, συγχαρητήρια στην εισηγήτρια που έκανε ε, τεράστιο έργο για να μπορέσει να εξετάσει όλες αυτές τις τροπολογίες και να αντιμετωπίσει πολύ δύσκολα θέματα. Ένα από τα πιο δύσκολα θέματα σε αυτό το σχέδιο κανονισμού είναι η έννοια του προστατευόμενου πελάτη. Και καλωσορίζω την συζήτηση για αυτό το θέμα και τη συμπερίληψη των ευάλωτων ε, πελατών ανάμεσα στους προστατευόμενους πελάτες. Είναι χρήσιμη αυτή η διαφοροποίηση και σύμφωνη με το ενδιαφέρον αυτής της Επιτροπής για την προστασία του καταναλωτή. Βεβαίως υπάρχει υποστήριξη και για τις συμβιβαστικέ τροπολογίες, αλλά θα πρέπει μάλλον να σας προειδοποιήσω για την δυσκολία που υπάρχει όσον αφορά το θέμα των ενδείξεων τιμών. Σύμφωνα με τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, είναι ξεκάθαρο ότι περίπτωση κρίσης θα υπάρξει έλλειψη φυσικού αερίου και ότι ε, θα αντιδράσουν και τιμές σε αυτή την έλλειψη. Είναι θέμα προσφοράς και ζήτησης. Άρα λοιπόν, αν τα κρατημέλη, οι αρχές θέλουν να το ρυθμίσουν αυτό, πολύ σύντομα θα θα ξεπεράσουν τα τρόπο λειτουργία της, ευρωπαϊκής, της εσωτερικής αγοράς και βέβαια και τις δυνατότητες χορήγησης φυσικού αερίου, παροχής φυσικού αερίου. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε, είναι πολύ δύσκολο βέβαια το θέμα και επικίνδυνο το θέμα των τιμών, διότι λέμε ότι η σωστή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς που σημαίνει ότι έχουμε τις απαραίτητες υποδομές και πολλά αφορούν τις ανάγκες σε υποδομές είναι η καλύτερη εγγύηση για την ασφάλεια ανεφοδιασμού. Μια λειτουργούσα αγορά είναι η καλύτερη εγγύηση για την ε, ανεφοδιασμό. Γιατί σε περίπτωση κρίσης σε κάποιο τμήμα της Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει αρκετό φυσικό αέριο σε άλλα, τμήματα της... Ε, σε άλλα μέρη της Ευρωπαϊκή Ένωση για να βοηθηθούν αυτοί που χρειάζονται αέριο. Και έτσι πρέπει να λειτουργεί η εσωτερική αγορά. Και προσπαθούμε μέσω της φιλοσοφίας αυτού του κανονισμού να διασφαλίσουμε πως η αγορά θα λειτουργεί όσο γίνεται περισσότερο. Και μόνο σε ακραίε περιπτώσεις μέτρα που ξεπερνούν την ευρωπαϊκή, αγνοούν την εσωτερική αγορά θα μπορούν να ληφθούν. Να σας πω, τον Ιανουάριο όταν περάσαμε την κρίση του φυσικού αερίου, φυσικά υπήρξε αντίδραση για τις, τιμές, υπήρξε αύξηση στις τιμές, η αγορά όντως ανταποκρίθηκε στη ζήτηση φυσικού αερίου σε διάφορες περιοχές. Υπήρχε δηλαδή αύξηση της τιμής που ήταν λογική. Και αυτή η αύξηση διήρκησε ένα περιορισμένο διάστημα χρονικό και αν το δούμε ε, σε επιτήσιας βάσεις, ο αντίκτυπος ήταν ε, αμεληταίος. Είναι επικίνδυνο παιχνίδι το να παίξουμε με τις τιμές, αν θέλουμε η εσωτερική αγορά να παίξει το ρόλο της και να έχουμε ασφάλεια ανεφοδιασμού. Εδώ λοιπόν ε, βάζουμε ένα ερωτηματικό στις σχετικές τροπολογίες, επιπλέον έχουμε επιφυλάξεις για τις τροπολογίες που προσπαθούν να δημιουργήσουν νέες αρμοδιότητες για θεσμούς που έχουν δημιουργηθεί από το τρίτο πακέτο εσωτερικής αγοράς όπως η ENSOC, δηλαδή το δίκτυο ε, των ε, φορέων συστημάτων μετά, μετάδοσης ή διάδοσης ή το νομάδα, το Συμβούλιο μάλλον ε, συνεργασίες για το φυσικό αέριο. Αυτοί οι θεσμοί δεν έχουν αρμοδιότητες, είναι βέβαια σημαντικά σώμα το πρέπει να τα διαβουλευόμαστε, αλλά δεν έχουν αρμοδιότητες για λήψη απόφασης και αυτό είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί. Και τέλος, αλληλεγγύη. Αλληλεγγύη είναι κάτι που πολύ σωστά είπε και ο κ. Σίβικ, είναι αμοιβαία αρμοδιότητα, ε, μάλλον ευθύνη των κρατών μελών και γι' αυτό και θέλουμε τα κράτη-μέλη και όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορεί, δηλαδή οι ρυθμιστικές αρχές, οι ε, αρμόδιοι για τα συστήματα ε, μεταφορά κτλ. Και όλοι όσοι ενδιαφέρονται να συνεργαστούν ώστε να έχουμε τα καλύτερα δυνατά μέσα για να αντιμετωπίσουμε του κίνδυνου που μπορεί να εντοπιστούν σε περίπτωση διακοπής της παροχής ε, ή προβλήματος στην παροχή. Να υπάρχουν δηλαδή σχέδια επίγουσας ε, ανάγκης, να υπάρχουν ε, σχέδια πρόβλεψης και εδώ είναι απαραίτητη η συνεργασία. Και στη συζήτηση που κάνω αυτή τη στιγμή με τα κρατημέλη, το στοιχείο αυτό λαμβάνεται υπόψη και πιστεύω πως το Κοινοβούλιο επίσης τονίζει την ανάγκη περισσότερη ελληνική που θα πρέπει να πάρει τη μορφή της περιφερειακής συνεργασίας στον σχεδιασμό προληπτικών πλάνων και πλάνων επίγουσας ανάγκης. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας και θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Καλνιέτε για να μας κάνει τις τελικές της παρατηρήσεις. Δεν άκουγα ε, εκείνη τη στιγμή. Συγγνώμη, κυρία Πρόεδρε. Θα, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή για τις παρατηρήσεις που έκανε και επίσης θα ήθελα να τονίσω την λέξη υπερβολική άνοδος των τιμών που θεωρώ ότι δεν ε, αντιστοιχεί προς τους πραγματικούς ε, μηχανισμούς διαμόρφωσης των τιμών. Είναι πολύ κοντόφθαλμη. Επίσης θα ήθελα να εκφράσω την ε, λύπη μου που ορισμένες από τις τροπολογίες δεν εμπέπτουν ακριβώς στην αρμοδιότητα της ΣΥΜΚΟ. Και όπως είπα θα τις ακολουθήσω και θα ήθελα να ενθαρρύνω τα μέλη της Επιτροπής ΣΥΜΚΟ να τις ε, καταθέσουν, εάν επιμένουν ότι είναι σημαντικές. Και αν κατακλείδη θα ήθελα να πω ότι αρχίζουμε την εργασία μας αυτό τον ε, ειδικό τομέα της ασφάλειας εφοδιασμού με, το με φυσικό αέριο σαν τμήμα κοινή ενεργειακής πολιτικής η οποία μόλις τώρα, ε, η οποία βρίσκεται εδώ και Και θα ήθελα να επενθυμίζω τις φιλοδοξίες που εξέφρασε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο οποίος ε, λέει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να διαματήσει αυτό το ρόλο, δηλαδή να διευκολύνει και να προαγάγει τη δημιουργία μιας φιλόδοξης κοινής, ε, μακρόπνοης κοινή ενεργειακής πολιτικής. Περισσότερο από όσα ε, που υπερβαίνει αυτό που υπάρχει στην παρούσα φάση. Ε, θα περιμένουμε λοιπόν τις μελλοντικές εξελίξεις και τους νέους ε, κανονισμούς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ. Perfetto, grazie mille, ringrazio. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ εσάς και όλους τους κέντρους συζητητές, καθώς και όσους συνέβαλαν ε, στη σύνταξη αυτής της έκθεσης με τις διάφορες τροπολογίες. Να θυμίσω ότι αύριο θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή στις 10 και 20, δηλαδή μετά από την ψηφοφορία που σας ανέφερα. Η ψηφοφορία στην Ολομέλεια θα γίνει το Φεβρουάριο. Και θα περάσουμε τώρα στο τελευταίο θέμα που έχουμε στην ημερήσια διάταξη και που συνδέεται με την ενημέρωση των καταναλωτών για τα τρόφιμα. Και θα δώσω το λόγο την κυρία Σέλντε Μόζε, την εισηγήτρια. Vi venter til et enkelt minut, imens folk forlader lokalet, så der bliver ro. Sì, direi di aspettare qualche minuto. Anche perché siamo molto in anticipo sui... Ναι, και γιατί έχουμε... πάει πολύ γρήγορα. Έχουμε πάει πολύ γρήγορα. Ja, jeg tror, jeg prøver stille og roligt. Penso che la situazione sia più tranquilla, quindi... Νομίζω πως κάπως ησυχάσαμε, οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε. Tak for det, fru formand. Jeg forsøger stille. Tak. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να ξεκινήσω. Ωρες ώρες υπάρχουν πολλές νομοθετικές προσπάθειες και πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί χρειάζεται να ασχολούμαστε με ε, τα θέματα των τροφίμων Εχθές λοιπόν μου, μου θύμισαν πόσο σημαντικό είναι να ε, προσπαθήσουμε να καταρτήσουμε σωστή νομοθεσία σε αυτό το τομέα. Παραδείγματος χάρη, ε, πάτε για παράδειγμα το διαβήτη. Έχουμε 30 εκατομμύρια Ευρωπαίους που πάσχουν από διαβήτη ή ε, έναν σημαντικότατο αριθμό θανάτων από διαβήτη κάθε χρόνο στην Ευρώπη, ο οποίος είναι εκπληκτικός. Ξέρω ότι 90% των ανθρώπων που πάσχουν από διαβήτη ε, πάσχουν από διαβήτη δευτέρου τύπου και στον διαβήτη δευκέρου τύπου πρόκειται για μια ασθένεια η οποία είναι ε, την οποία μπορούμε να προλάβουμε και να μπορέσουμε να επιτρέψουμε στα άτομα αυτά να ζήσουν μια φυσιολογική ε, ζωή. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε σωστές πληροφορίες για τους καταναλωτές σχετικά με τα τρόφιμα για να μπορούν να λαμβάνουν τις σωστές τους αποφάσεις. Βεβαίως, θα πρέπει αυτό να αναφερθεί και ε, από πλευράς βιομηχανικής, αλλά το πιο βασικό είναι ε, πώς θα υποφεληθούν οι ε, πολίτες οι οποίοι αγοράζουν αυτά τα προϊόντα. Δεν μπορώ να πω ότι θα εξαλείψουμε το διαβήτη στην Ευρώπη, αλλά η νομοθεσία μπορεί να συμβάλλει να υπερβούμε αυτό το γεγονός στην Ευρώπη και γι' αυτό πρέπει να κάνουμε το, την προσπάθεια να γίνει σωστή ε, νομοθεσία. Η Επιτροπή μας η οποία έχει ε, την ε, ηγεσία σε αυτό το θέμα έχει διατυπώσει 210 τροπολογίες και ο Μάικ Ταραμπέλα στην Επιτροπή Γεωργίας έχει διατυπώσει 83 τροπολογίες. Εμείς έχουμε ε, μόνο 80. Και αυτό πριν αρχίσει η Ολομέλεια να υποβάλει ε, τροπολογίες. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι διαφαίνεται μία σοβαρή μάχη, αλλά πρέπει να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας για να μπορέσουμε να καταλήξουμε υπό την ηγεσία της Επιτροπής Περιβάλλοντος ε, που ε, ε, έχει αναλάβει την έκθεση αυτή κατά πρώτον λόγων, να έχουμε μία συνεκτική λύση. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι οι, υπόλοιπες, ε, οι περισσότερες τροπολογίες τις οποίες αναφέρω είναι τροπολογίες οι οποίες ε, είχαν ήδη διατυπωθεί την άνοιξη. Δηλαδή οι περισσότερες τροπολογίες προέρχονται από την πλειοψηφία την οποία είχαμε ψηφίσει την Άνοιξη. Και αυτό θα πρέπει να γνωρίζετε καταρχήν προτού εξετάσετε τις προτάσεις μου. Εγώ όμως αποφάσισα να επικεντρωθώ σε τρεις τομείς ε, ε, όπου το θέμα διαφέρει από τις προτάσεις που είχαν διατυπωθεί την Άνοιξη όπου λέγαμε ότι πρέπει να υπάρξει μία συνολική εξαίρεση για τα αλκοολούχα ποτά ενώ εγώ προτείνω όλα τα αλκοολούχα πρώτα να περιληφθούν σε αυτή την ε, οδηγία. Ίσως είναι αντιφατικό, αλλά πιστεύω ότι είναι βασικό να το συζητήσουμε διότι ε, το ενόπνευμα μπορεί να είναι και ένα πολιτιστικό πρόβλημα και επηρεάζει πάρα πολύ την υγεία μας. Γι' αυτό και ίσως θα έπρεπε να ενημερώσουμε τους καταναλωτές για το περιεχόμενο όλων των υνοπνευματοδών ε, ποτών που περιλαμβάνουν ε, διάφορες ουσίες πολυβραβερές. Εγώ σαν ε, καταναλωτής και πολίτης θα ήθελα να τα γνωρίζω όλα αυτά παρόλο που από καιρού καιρών πίνω ένα ποτηράκι. Η διαφορά με σε σχέση με την προηγούμενη έκθεση είναι ότι αναφερόμαστε εδώ ή στη σηματοδότηση. Και ε, υπάρχουν διάφορες ε, δυνατότητες, πρέπει όμως να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τους καταναλωτές να διαβάζουν το περιεχόμενο. Θα μπορούσαμε να είχαμε δηλαδή το σύστημα με τους κωδικούς και εγώ σε αυτό αναφέρομαι. Θα ήθελα όμως να σας θέσω το θέμα για να μπορούμε όλοι να γνωρίζουμε τι είναι εύκολο. Δηλαδή τι θα βοηθήσει τους καταναλωτές να καταλάβουν καλύτερα όλες τις πληροφορίες που περιέχει η σήμανση. Θα χρειαστεί λοιπόν μια κωδικοποίηση. Επιπλέον πιστεύω ότι η συσκευασία θα πρέπει να αναφέρεται εις ε, την συνολική ενέργεια η οποία περιλαμβάνεται σε κάθε προϊόν και αυτό θα πρέπει να αναφέρεται στο μπροστινό μέρος της ε, συσκευασίας, δηλαδή ποιο είναι το ενεργειακό περιεχόμενο του περιεχομένου, αλλά εγώ θα έλεγα ε, μπροστά να αναφέρουμε τις, ε, τις ε, θερμίδες ανά 100 γραμμάρια με χρώματα γιατί αυτό έχει αποδειχθεί ότι διευκολύνει την κατανόηση των καταναλωτών και ιδιαιτέρως είναι εύκολο για τους καταναλωτές όταν συνδυάζουμε τους αριθμούς ε, με τα χρώματα για να είναι εύκολο να διαβάσουν αυτές τις πληροφορίες. Όσον αφορά την τρίτη συγκεκριμένη πρόταση που θα ήθελα να διατυπώσω, είναι ότι συνιστώ να να αναφέρουμε την ε, συνιστόμενη ε, ημερήσια περιεκτικότητα η οποία δεν πρέπει να είναι το επίκεντρο ε, των πληροφοριών που θα δίνονται για κάποιο προϊόν και εδώ αναφέρομαι στις γενικές μου προτάσεις μόνο. Θα ήθελα όμως να σας ρωτήσω πώς θα έπρεπε να ξεκινήσει η συζήτηση όσον αφορά το μέγεθος των συσκευασιών διότι το πρόβλημα είναι το εξής. Υπάρχουν ορισμένα ε, τρόφιμα τα οποία διατίθενται μόνο σε πολύ μικρές συσκευασίες και θα πρέπει να αλλάξει η συσκευασία τους, να μεγαλώσει κάπως, διότι ε, αυτό θα διευκολύνει και ε, δεν θα χρειάζονται πλέον τόσες πολλές πληροφορίες και ε, ε, εάν είναι μικρός ο χώρος θα είναι πολύ δύσκολο να διαβάσει κανείς την ετικέτα. Εδώ λοιπόν τίθεται ένα ερώτημα το οποίο να απευθύνω προς την Ομίγυρη. Έχω ακόμη δύο παρατηρήσεις και μετά θα ολοκληρώσω. Ε, η ημερομηνία για τις τροπολογίες είναι 7 Ιανουαρίου, μάλλον 6 Ιανουαρίου. Λάθος, 11 Ιανουαρίου. Εν... Με συγχωρείτε. Ίσως λάθος διάβασα. Νόμιζα ότι ήταν 6 Ιανουαρίου, αλλά φαίνεται ότι έχει μετατεθεί στις 11 Ιανουαρίου και ε, ελπίζω ότι θα ξανασυναντηθούμε τώρα μετά τις χριστουγεννιάτικες διακοπές μας. Αυτό ήταν το ένα σχόλιο και το άλλο είναι ότι στην επόμενη εβδομάδα του Στρασβούργου θα συγκαλέσω τους συζητητές για να συζητήσουμε ε, το θέμα και να δούμε αν μπορούμε να προσεγγίσουμε τις θέσεις μας προτού ξεκινήσουμε να διαπραγματευόμαστε τις ε, τροπολογίες και να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Είναι πολύ βασικό βέβαια να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια συμβιβαστική λύση η οποία να ικανοποιεί όλους παρόλο που έχω συγκεκριμένα σκέψη επί του θέματος και αυτό ήταν σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Να δώσω το λόγο στη Σκιώδη. Εισηγείται την κυρία Κοράτσα Βίλτ. Ευχαριστώ, Λάρα. Να ξεκινήσω λέγοντας πόσο πολύ καλή ήταν η συνεργασία με την ε, εισηγήτρια. Και είμαι σίγουρη ότι θα τα καταφέρουμε να βρούμε η θέση. Πραγματικά εκτιμώ τα ενέκθεσή σας και συμφωνώ σε πολλά θέματα. Να ξεκινήσω λέγοντα ποια είναι η αρχή ή ποιο είναι το όραμα από το οποίο προέρχονται τα σχολεία μας. Θα πρέπει να δώσουμε ε, δύναμη και να όθησε στον καταναλωτή. Δεν είναι ένα παθητικό παιδί, είναι ένα άνθρωπο που έχει πλήρε ευθύνε και θα πρέπει από εμά του πολιτικού να του δοθεί η ευκαιρία να κάνει την καλύτερη δυνατή ενημερωμένη επιλογή. Θα πρέπει να ενημερώνουμε και να εκπαιδεύουμε, όχι να επηρεάζουμε, να αποφασίζουμε για τον καταναλωτή. Σας ευχαριστώ. Αυτή είναι μια βασική αρχή που εξαιρετικά σημαντική Δηλαδή να δώσουμε στον καταναλωτή περισσότερα μέσα ώστε να μπορεί να έχει ελεύθερη επιλογή. Η άλλη, ο άλλος πυλώνας είναι η ελεύθερη αγορά, κατά την απόψή μου. Εγώ είμαι κατά οποιοδήποτε μέτρου που θα παρεμπόδιζε την ορθή λειτουργία και την ελεύθερη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, διότι, όπως πολλοί από σας συμφωνείτε εδώ, είναι η ελεύθερη αγορά ε, και ε, ωφέλιμη για όλους, για τις εταιρείε, για τον καταναλωτή, για όλους. Γι' αυτό και είμαι κατά του φαναριού, γιατί αυτό είναι ο τρόπο να πούμε στον καταναλωτή: Εγώ ξέρω ποιο είναι το καλύτερο για την υγεία σου. Αντί να του πούμε ότι έτσι έχει κατάσταση αντικειμενικά και μπορεί τώρα να διαλέξει από μόνο σου. Κάτι άλλο είναι για το θετικό σύστημα διατροφής. Είναι η ίδια αντίληψη. Τι είναι η καλή υγεία. Μπορεί κανείς να πει και να είναι πολύ ξεκάθαρος ποια πράγματα απειλούν την υγεία, ποια είναι ζημιογόνα για την υγεία, γιατί αυτά θα πρέπει να απαγορεύονται. Αλλά όλα τα υπόλοιπα μπορεί να είναι πολύ υγιές για ένα παιδί, να καταναλώνει πολύ ε, λίπος. Είναι πολύ κακό να τρως βούτυρο από την άλλη άμα είσαι χολυστερίνη. Δεν είναι εύκολο να τα βάλουμε όλα σε ένα ε, καλούπι. Ο καταναλωτής είναι παιδιά, ενήλικες, γυναίκες, άντρες, ε, γέροι, νέοι, υγιείς άνθρωποι, άνθρωποι που ζυγίζουν 40 κιλά, άνθρωποι που ζυγίζουν 80 είναι πολύ μεγάλη διαφορά για το πόσο λίπος, πόσο αλάτι και πόση ζάχαρη μπορεί να καταναλώνουν. Μπορώ να σας πω ότι το λίπος στο τυρί παρμεζάνα είναι πάρα πολύ υγιές, ακόμα και βάζουν στη συσκευασία 32% λιπαρά και ο κόσμος τρομάζει. Είναι απλά ένα παράδειγμα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι το λίπος είναι πάντα ανθυγινό και η ζάχαρη είναι πάντα ανθυγινή. Τα παιδιά χρειάζονται περισσότερη ε, ζάχαρη από ότι οι ενήλικες. Είμαι κατά λοιπόν όλων αυτών των συμβόλων και κατά της υποχρεωτικής υποχρεωτικού της υποχρεωτικής αναγραφής της ε, ημερήσιας δόσης. Γιατί πώς μπορεί να ξέρει κάθε τι είναι καλό για μένα, για το παιδί μου που είναι πέντε χρονών, ενώ για σένα, ας πούμε, που είσαι ένας ε, γερός υγιής άνδρας, ποια είναι η σωστή ημερήσια δόση. Να ενημερώνουμε τον καταναλωτή και όχι να το επιβάλλουμε. Αν και προέρχομαι από τον βόρειο κόσμο, η τροφή και τα αλκοολούχα ποτά, ακόμα και τα μεικτά προϊόντα, δεν είναι τα ίδια. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να ρυθμιστούν. Λέω ότι θα πρέπει να ρυθμίζονται με διαφορετικό τρόπο και είναι αλήθεια πως ε, τα αλκοολούχα ποτά έχουν ε, θερμίδες και θα πρέπει και αυτό να το λάβουμε υπόψη. Αλλά υπάρχει ήδη οδηγία για το κρασί και θα έπρεπε ίσως να δούμε να το δούμε και να το ρυθμίσουμε με χωριστό τρόπο, αλλά όχι μαζί με τα τρόφιμα. το μέγεθος είναι πολύ σημαντικό και όχι μόνο το μέγεθος, αλλά και το χρώμα, η αντίθεση, αλλά τελικά να σας πω ότι εκνευρίζομαι πολύ αν πάω στις 7 η ώρα το βράδυ σε μια Παρασκευή. Δεν έχω τα γελιά μου μαζί, γιατί μια γυναίκα άνω το 40 δεν θα πρέπει να αγωνίζεται με ένα πακέτο για 10 λεπτά, ενώ το παιδί της ουρλιάζει δίπλα της για να δει ποια είναι τα βασικά συστατικά για να κάνει την επιλογή της. Άρα λοιπόν πρέπει να είναι όλα αυτά ευανάγνωστα, απλοποιημένα. Λένε και χτυπιούνται και οδύρονται στην Επιτροπή Περιβάλλοντος ότι πρέπει όλα να αναγράφονται στο πακέτο στη συσκευασία. Πρέπει να υπάρχει καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην ενημέρωση και στη συσκευασία. Δεν χρειάζεται όλο το πακέτο να είναι αφιερωμένο στη διαφήμιση για να έχει το Spider-Man, ας πούμε, πάνω. Θα πρέπει να απολοποιήσουμε, λοιπόν, να γίνουν όλα τόσο όσο γίνεται πιο κατανοητά. Αλλά τι καταλαβαίνει ο κόσμος και όχι και όχι νάτριο. Άρα αυτό που θα πρέπει να γράφει απάνω στη συσκευασία θα πρέπει να λέει αλάτι τόσο στους πίνακες. Να υπάρχει ένα πίνακα όπου βάζουν, μπαίνουν όλα αυτά. Επιλογή, προαιρετική, μυρίσια μερίδα, ε, θερμίδες κτλ. Όσο περισσότερα μπουν στο μπροστινό κομμάτι του πακέτου, τόσο λιγότερα καταλαβαίνει ο καταναλωτής. Ε, τώρα, για τις αλλεργίες, Αλλεργίες ε, Δύο φορέ έχω πάει στο νοσοκομείο γιατί έχω ένα πεντάχρονο παιδάκι που είναι πολύ αλλεργικό και δεν θέλω άλλοι γονεί να περάσουν τα ίδια. Άρα λοιπόν πληροφορίε για τις αλλεργίες που απελούν τη ζωή και για τέτοια συστατικά θα πρέπει να είναι ευανάγνωστα. Και με έχω βαρεθεί με αυτή τη σημείωση που λέει ότι μπορεί να υπάρχουν ε, ίχνη ξηρών καρπών. Υπάρχουν ή δεν υπάρχουν υπάρχουν και, ή δεν υπάρχουν, που είναι κακό για τον καταναλωτή. Ε, πραγματικά με ενδιαφέρει αυτό το θέμα, όπως καταλαβαίνετε, και το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι είμαι υπέρ κάθε δυνατής προσπάθειας για να υπάρξει εναρμονισμένη προσέγγιση. Είμαι κατά της πρότασης της Κομισιόν να αφήσουμε τα κράτη-μέλη ε, να διαλέξουν ε, και να κάνουν διαφορετικούς εθνικούς κανονισμούς, γιατί αυτό θα ήταν εμπόδιο στην εσωτερική αγορά και θα προκαλούσε σύγχυση στον καταναλωτή. Και φυσικά όταν ε, μπαίνει ένα προϊόν στην ευελική αγορά θα πρέπει να μπορεί να μπει και στην υπόλοιπη αγορά. Όσο γίνεται πιο εναρμονισμένα, τόσο το καλύτερο για τον καταναλωτή και για την εσωτερική αγορά. Αυτές είναι αρχικές μου ε, παρατηρήσεις. Ευχαριστώ Λάουρα. Σας ευχαριστώ για την παρέμβαση. Θα δώσω τώρα το λόγο στον Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Α, αυτές τις μέρες άκουσα μια διάλεξη όπου ένας καθηγητής, έλεγε ότι η αναφορά της θρεπτικής αξίας ε, δεν παίζει ρόλο. Σημασία έχει η σύνθεση των θερμίδων ανά ημέρα. Ε, τότε μπορούμε να συζητήσουμε κατά πόσο όλη αυτή η οδηγία είναι αναγκαία. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω μαζί σας ε, ότι εάν ε, κάνουμε μία οδηγία δεν χρειάζεται να υπάρχουν πολλά, δεν πρέπει να υπάρχουν πολλά περιθώρια ερμηνείας, γιατί τότε έχουμε να διευκρινίσουμε καταρχήν την ίδια την οδηγία και μετά τους ε, επιμέρους κανονισμούς της χώρες ε, μέλης, μέλη. Και αυτό ενισχύει την ε, γραφειοκρατία και δεν νομίζω ότι έχει απολύτως κανένα πλεονέκτημα για τον καταναλωτή, ούτε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να επισέλθω τώρα σε ορισμένα στοιχεία της έκθεσης της κυρίας Σαλντεμόζε. Θέλουμε έναν όριμο καταναλωτή, όχι έναν υποκειδεμόνευση καταναλωτή. Θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ο καταναλωτής θα πρέπει όταν πηγαίνει στο ράφι του σούπερ μάρκετ να έχει δυνατόν σύντομες και επαρκείς πληροφορίες, όχι υπερβολικά πολλές, γιατί θα πρέπει να πάρει μια απόφαση και όταν τον σκοτώνουν οι πληροφορίες είναι δύσκολο να πάρει μια απόφαση μπροστά στο ράφι. Γι' αυτό ε, βεβαίως έχει νόημα να έχουμε ενίες ε, ενιαία σήμανση. Ε, για παράδειγμα τα 100 γραμμάρια, τα 100 μιλιγκράμμ για να έχει τη δυνατότητα σύγκρισης καθώς και την μερίσια δόση ενδεχομένω Μπορεί αυτό να γίνεται εκουσίωσο. Το ερώτημα είναι ε, τι λένε τα 100 γραμμάρια ή τα 100 μιλιγκράμμ. Ε, δεν ξέρω εάν μια βιομηχανία που παράγει τσίχλες λέει ότι η μερίσια δόση είναι δεν ξέρω πόσες τσίχλες, ε, όλα αυτά μας οδηγούν ενδεχομένω σε παραλογισμούς. Τώρα, όσον αφορά το κρασί, και εδώ είμαι ιδιαίτερως επιφυλακτικός, γιατί στη Γερμανία είναι, ε, ανήκει και στην πολιτική μας ε, και στην παράδοσή μας και ενδεχομένως ε, ευνοεί, βοηθάει και την υγεία. Τώρα, ε, δεν ξέρω τι βοηθάει η αναγραφή σε θερμίδες, περιεκτικότητας του κρασιού σε θερμίδες. δεν νομίζω ότι θα πρέπει να αλλάξει πάρα πολλά πράγματα όσον αφορά τα αλκοολούχα ποτά. Η έκθεση κ. Φαλτεμόζε ε, προβλέπει να εξαιρεθούν τα αλκοολούχα ποτά. Είπατε ήδη ότι υπάρχει μια σχετική οδηγία εντό οποία μπορεί να ρυθμιστεί το θέμα των, των αλκοολούχων ποτών. Τώρα, όσον αφορά την αναφορά της χώρας προέλευσης, εδώ θα πρέπει να ξέρουμε ότι δημιουργείται με τον τρόπο αυτό μια τεράστια γραφειοκρατία. Πώς θέλετε να παρακολουθήσετε όλα αυτά, πώς θέλετε να ορίσετε όλα αυτά. Γι' αυτό θα πρέπει να έχετε κατά νου όταν θέλετε να θεσπίσετε τις διατάξεις, ότι εκείνοι που καλούνται να τις στηρίσουν, ε, όλα αυτά συνδέονται με κόστος, με τη δημιουργία γραφειοκρατίας και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις τελικά επιβαρύνονται πολύ περισσότερο με αυτό το επιπρόσθετο κόστος, πολύ λιγότερο οι μεγάλες επιχειρήσεις. Γι' αυτό έχει νόημα να σκεφτούμε ότι θα πρέπει όλα αυτά να ελαχιστοποιηθούν ή δυνατόν. Θα πρέπει να υπάρχει μια ξεκάθαρη αναγνωσιμότητα των στοιχείων αυτών και βεβαίως εδώ γνωρίζουμε ότι δημιουργούνται προβλήματα. Τα τρία χιλιοστά της Επιτροπής. Ε, για να επιτευχθεί αυτό χρειάζονται δράσεις συσκευασίε. Η κ. προτείνει 1,2 χιλιοστά, αλλά οι συσκευασίε θα πρέπει να είναι εύχρηστες Γι' αυτό θα πρέπει, νομίζω, να διδικωθεί ω εξή. Θα πρέπει να είναι καθαρά ευανάγνωστο και θα πρέπει να υπάρχει ένα περιθώριο ευελιξία όσον αφορά το μέγεθο του προϊόντο. Δηλαδή, η συσκευασία για τι τσίχλε ε, είναι διαφορετική από τη συσκευασία για τα τσίψε. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν και ένα περιθώριο ευελιξία σε σχέση με το μέγεθο του προϊόντο. Ε, δεν θα πω άλλα πράγματα. Θα μπούμε στι λεπτομέρειε κάποια άλλη στιγμή αλλά η θερμή μας παράκληση είναι να περιλαμβάνονται τόσες πληροφορίες στη σήμανση που να είναι εύπεπτες, να μπορεί να τις αφομοιώσει μάλλον ο καταναλωτής και να μπορεί να τις λάβει υπόψη του για να πάρει μια απόφαση. Δεν θα πρέπει να σκοτώνουμε τον καταναλωτή με υπερβολικά πολλές πληροφορίες γιατί στην περίπτωση αυτή ε, πετυχαίνουμε το αντίθετο και δεν μπορεί αυτό να είναι εις του καταναλωτού. Ε, Επίση για τις μικρομεσαίες επιχείρησεις, όπως σας είπα, όλα αυτά συνεπάγονται ένα επιπλέον κόστο. Και όταν θα σπίσουμε οδηγίε, θα πρέπει οι οδηγίε αυτέ να είναι δεσμευτικέ. Γιατί αλλιώ αυξάνουν τη γραφειοκρατία και οι επιχειρηματίες δεν γνωρίζουν ποιες διατάξεις θα πρέπει να τηρούν σε ποια χώρα και όλα αυτά δεν οδηγούν σε μια μεγαλύτερη εναρμόνιση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας. Ε, το λόγο έχει η κυρία Ρούλε. Ευχαριστώ. Τώρα <clears throat> θα μιλήσω εν ονόματι της Εμιλή Τούριν που δεν παρίσταται σήμερα. Σας ευχαριστώ για την καλή συνεργασία ε, με την κυρία Σάρντε Μόζερ. Έχει, ε, μου έχει δώσει ένα σημείωμα αλλά θα αποκλίνω γιατί βλέπω ότι οι συνάδελφοι ε, παρουσιάζουν διαφορετικά το θέμα και έτσι πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε στους καταναλωτές ε, τις σωστές πληροφορίες που δεν έχουν πάντοτε. Θυμάμαι όταν ήμουν παιδιά όταν ήταν μικρά τα παιδιά μου υπήρχε ένα πρόβλημα για το παιδικό τσάι και ουσιαστικά αρρώστεναν τα παιδιά λόγω του ποσοστού ζάχαρης που είχε το παιδικό τσάι και ο καταναλωτής πρέπει να έχει τις πληροφορίες που χρειάζεται. Πρέπει να είναι απλές πληροφορίες, συμφωνώ, κατανοητές, αλλά είναι εύκολο να έχει κανείς κατανοητές πληροφορίες. Όταν λοιπόν θέλουμε να προσεγγίσουμε το καταναλωτή και να του δώσουμε ε, ακριβώς τις πληροφορίες, είναι εύκολο να το κάνουμε ε, και να ικανοποιήσουμε τον καταναλωτή. Μετά, το ενόπνευμα. Συμφωνώ και εγώ δεν θα ήθελα να προσθέσω πολλές πληροφορίες στις ετικέτες του κρασιού, αλλά το ινοπνεύμα έχει πολλές θερμίδες και δεν το ξέρουν όλοι. Ε, πολλοί δεν γνωρίζουν πόσο είναι το ποσοστό των θερμίδων του ινοπνεύματος και καλό θα ήταν να τους το πούμε. Αντί να τους επιβαρύσουμε με άλλες νομοθεσίες. Ε, επίσης για τη βιομηχανία. Όλα θα πρέπει να παρουσιάζονται σε ένα σημείο. Ε, πρέπει να προσπαθήσουμε να ε, παρουσιάσουμε τα πάντα κατά τρόπον ικανοποιητικό για τον καταναλωτή και τον πολίτη. Θεωρώ ότι οι ιδέες σας είναι καλές, κυρία Σαλτεμόζαρα, αλλά δεν μπορώ να συμφωνήσω σε όλα τα οποία είπατε. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Γκουζούσνικ. Πανή Ψεσεράιτσι, μια τον nedá, abych to, Λοιπόν, ε, και εμένα τα σχόλιά μου ακολουθούν την ίδια σκέψη όπως και των προηγουμένων δεν έχω παρακολουθήσει συνεδρίαση από την αρχή γιατί είμαι στην αντιπροσωπεία της Ονδούρας και γι' αυτό με πιέζει ο χρόνος. Ε, νομίζω όμως ότι εδώ το θέμα ε, δεν είναι πολύ περίπλοκο και πιστεύω ότι ο καθένας μπορεί να εκφραστεί. Εγώ πρέπει όμως να σας πω ότι δεν καταλαβαίνω καθόλου γιατί τσακωνόμαστε εδώ. Όταν δηλαδή σας ε, ακούω όταν ε, ακούω για το μέγεθος των ε, γραμμάτων, ε, τα χρώματα, τις ετικέτες, τη σήμανση για τις αλλεργίες, για τις ουσίες, Ε, δεν θα έπρεπε οι ψηφοφόροι μας να έχουν όσες πληροφορίες έχουμε κι εμείς. Και πιστεύω ότι ο καταναλωτής δεν είναι ανόητος θα μπορέσει να προσαρμοστεί. Δεν πρέπει δηλαδή εδώ να υποκαταστήσουμε τον καταναλωτή, αλλά να αποφύγουμε τη γραφειοκρατία και να εξοικονομήσουμε χρήματα στον καταναλωτή. Ε, αυτή είναι η πολιτική μου διακήρυξη και ευχαριστώ το γεγονός που ανέφερε η συνάδελφος Έμα και το οποίο θα σας παρουσιάσει στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ. Le, le lascio ora la parola alla signora Wengsberg. Ε, Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε που περιμένατε να έρθω στη θέση μου. Θα πρέπει να σας πω ότι χαιρετίζω τη σήμανση των τροφίμων ως τον ενδεδειγμένο τρόπο για να ενημερώνονται οι καταναλωτές. Αλλά ε, έχω επίσης την άποψη ότι η σήμανση των τροφίμων από μόνη της δεν επαρκεί και χρειαζόμαστε για παράδειγμα μια ενημερωτική εκστρατεία, μια εκπαίδευση με τη διατροφή εν γέννη. Ωστόσο είμαι υπέρ αυτής της πρότασης και είμαι υπέρ της ενημέρωσης των καταναλωτών. Το ερώτημα είναι πώς θα πρέπει να γίνεται αυτή η ενημέρωση. Κατά βάση θα πρέπει να πω και η συνάδελφος ε, ε, ανέφερε κάποιες ε, εξαιρέσεις σχέση με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εγώ θεωρώ ότι για τις μεγάλες βιομηχανίες, για τους μεγάλους ομίλους, την κράφτια για παράδειγμα, μπορούμε να απαιτήσουμε ορισμένα πράγματα, αλλά θα πρέπει να προσέξουμε τα πράγματα αυτά να είναι εφαρμόσιμα στην πράξη και χρειαζόμαστε κάποιες εξαιρέσεις για τις μικρές επιχειρήσεις όπως είναι οι φούρνοι ή τα κρεοπολία που έχουν κάποιες μικρές συσκευασίε, ε, μικρής κλίμακας. Όσον αφορά τη σήμανση για τις αλλεργίες, για τους αλλεργιογόνους παράγοντες, νομίζω ότι εδώ η κυρία Ζόμαρα έκανε μια πολύ καλή πρόταση, ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ε, ε, υπάρχει ήδη μια σήμανση, αλλά θα πρέπει να προσέξουμε όσον αφορά τις μικρές επιχειρήσεις ε, για τα μη προσυσκευασμένα τρόφιμα. Θα ήθελα να τονίσω κάτι στο οποίο νομίζω ότι μπορούμε να πετύχουμε ομοφωνία. Το έθεσα και την περασμένη φορά. Έχω την άποψη στην προστινή πλευρά, όπως προτείνει και η κυρία Ζόμερ της συσκευασία, θα πρέπει οι κατασκευαστές να υποχρεώνονται να έχουν μία σήμανση εάν αντί, αν χρησιμοποιούν να διατηρεί ένα άλλο συστατικό για τα υποκατάστατα. Θα πρέπει να υπάρχει μια ειδική σήμανση. Και θα ήθελα να πω ότι είχαμε θετικές αντιδράσεις, για παράδειγμα, από τη γαλακτοβιομηχανία. Ε, νομίζω ότι είναι επιθυμητή η συνεργασία τους και νομίζω ότι τώρα που βρισκόμαστε στη φάση διατύπωσης των τροπολογιών θα πρέπει όλες οι πολιτικές ομάδες να συμφωνήσουν για αυτή την τροπολογία όσον αφορά την αντικατάσταση ορισμένων ουσιών ε, και θα με χαραπούσει πάρα πολύ η συνεργασία από όλες τις πολιτικές ομάδες. Τώρα, ένα θέμα που έχουμε διαφορετική άποψη. Ε, καταρχήν θα ήθελα να τονίσω το θέμα ε, στο οποίο συμφωνούμε όσον αφορά την ημερήσια δόση, το GDA. Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλό να την καταργήσουμε αναφερόμενη σε μία μεσαία τιμή. Ε, λέγοντας αναφερόμαστε σε μία μεσαία τιμή. Πώς ορίζουμε αυτή τη μεσαία τιμή. Ε, ε, την ποσοστιαία ημερήσια ανάγκη σε θερμίδες. δεν είναι δυνατόν, δεν μπορούμε παρά να έχουμε μια, έναν μέσο όρο της ημερήσιας ε, ανάγκη σε θερμίδες κατά μέσο όρο. Δεν μπορούμε να κάνουμε τη διάκριση σε διάφορες ομάδες, παιδιά, και κλπ. Εγώ προσωπικά ε, θεωρώ ότι θα έπρεπε να αναφέρουμε μόνο τις θερμίδες, γιατί αν αναφέρουμε την περιεκτικότητα σε λίπος κλπ, θεωρώ ότι οι πληροφορίες αυτές είναι άχρηστες. Εγώ είμαι υπέρ του GDA, δηλαδή τη ημερήσία ανάγκης σε θερμίδες. Έτσι κι αλλιώς οι βιομηχανίες το κάνουν αυτό σε πολλούς τομείς. Αλλά θα πρέπει να προσέχουμε οι μεγάλες βιομηχανίες να μην ε, ε, έχουν διαφορετικά σημεία αναφοράς. Δηλαδή, ε, μια φορά να αναφέρονται σε 500 γραμμάρια, δηλαδή μισή πίτσα ή και σε κάποια άλλη συσκευασία να αναφέρονται στις ημερήσεις ανάγκες για 20 γραμμάρια γιατί αυτό οδηγεί σε κάποια σύγχυση. Τώρα, όσον αφορά τα φώτα σηματοδότησης. Νομίζω ότι αυτό οδηγεί σε παρανοήσεις και σε σφαλμένη διατροφή. Αν υπάρχει κόκκινη σήμανση σε ένα τρόφιμο, ο καταναλωτής ίσως θεωρεί ότι το προϊόν είναι βλαβερό. Ενώ ε, για παράδειγμα, ε, για μια ισορροπημένη διατροφή χρειάζεται κανείς ε, ενδεχομένως λίπος ή κάποιοι φυσική χημοί που έχουν την πράσινη σήμανση. Εγώ <laughs> θα ήθελα να σας πω το επιχείρημα, αν το μετρικό γάλα το συσκευάζαμε και βάλαζαμε μια σήμανση θα του βάζαμε κόκκινο. Συνεπώς λοιπόν θεωρώ ότι μπορεί να οδηγήσει σε παρανοήσεις η μέθοδος αυτή της σήμανση βάσει των σημάτων της ε, τροχέας, της κυκλοφορίας, κόκκινο ή πράσινο. Νομίζω ότι θα πρέπει κάπως να διευκρινίσουμε το θέμα του GDA, της ημερήσιας ε, ανάγκης στα ε, νομίζω ότι θα πρέπει να είναι εύληπτο από τον καταναλωτή εάν φάω αυτό το κομμάτι πίτσας, τότε θα έχω φάει ένα, ποσοστό, ένα ποσό λίπος, το οποίο αναλογεί στην τάδε ποσοστιαία ανάγκη μου σε λίπος. Στην ημερήσια δηλαδή. Σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Μάρτερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εν μέρη, υπόθηκαν τα όσα ήθελα να πω. Εν πάση περιπτώσει, εξ αρχής να πω ότι συμμερίζομαι τα όσα είπε η σκιώδη συζητήτρια και θέλω να πω να μιλήσω για το θέμα του φαναριού με μια άλλη οπτική. Δηλαδή να τονίσω την ανάγκη να υπάρξει κάποιο σημάδι που να βοηθά τον καταναλωτή να αποφασίσει. Το φανάρι είναι ένα ε, ένα σχέδιο, αλλά υπάρχουν και τα χρώματα με τα οποία μπορούμε να δώσουμε πληροφορία στον καταναλωτή. Εγώ δεν συμφωνώ με τη χρήση του φανάριου ακριβώς για αυτό το λόγο. Επειδή δηλαδή, όπως είπαν ήδη κάποιοι συνάδελφοι, το κόκκινο είναι αυτό στο οποίο σταματάμε, ενώ το πράσινο είναι αυτό που μας κάνει να προχωρήσουμε και το πορτοκαλί είναι το ενδιάμεσο, δηλαδή επέκειται κίνδυνος. Άρα λοιπόν εδώ εμείς θα, θα υποκαταστήσουμε τον καταναλωτή, θα δώσουμε ήδη μια ένδειξη να μην επιλέξει αυτό το προϊόν. Ακόμα περισσότερο αν αυτό είναι ένα σχέδιο με χρώμα, χρωματιστό. Όμως, επειδή πρέπει να βρούμε μία συμβαστική λύση, με φοβίζει το ότι εστιάζουμε την προσοχή στο φανάρι και να φτάσουμε να πούμε όχι για το φανάρι αλλά σβάλουμε το χρώμα γιατί θα πέσουμε στο ίδιο Λάθο. Η χρήση του κόκκινου, άσχετα από το αν θα χρησιμοποιήσουμε την εικόνα του φαναριού, είναι πάλι σήμα κινδύνου. Το κόκκινο σημαίνει κίνδυνος και ακριβώς γι' αυτό, εμεί αντίθετα, με ένα σχέδιο και με το χρώμα θέλουμε να δώσουμε μια πληροφορία στον καταναλωτή που μπορεί να μας θέσει σε να μας κάνει να τον υποκαταστήσουμε. Θα πρέπει λοιπόν να αποφύγουμε όχι μόνο το σήμα του φαναριού αλλά και τα χρώματα. Και θα κάνω μια πρόταση, μια πρόκληση αν θέλετε. Αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τα χρώματα, γιατί να μην χρησιμοποιήσουμε το μπλε για να πούμε ότι είναι ένα τρόφιμα που έχει, ένα τρόφιμα που έχει πολλές θερμίδες, το γκρι για ένα μεσαίο και το καφέ που έχει λίγες, θα διαπιστώσουμε αμέσως πως αυτά τα χρώματα δεν έχουν κανένα νόημα. Δεν ε, δείχνουν τίποτα στον καταναλωτή, δεν μεταδίδουν καμία πληροφορία. Άρα λοιπόν ε, αυτόματα σημαίνει αυτό πως δεχόμαστε το κόκκινο και το πράσινο, σημαίνει όχι στην αγορά, πράγμα το οποίο θα στρέβλουν την αγορά και δεν είναι αυτό που επιθυμούμε, ούτε είναι και προς το συμφέρον του καταναλωτή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει η κυρία Κέλλη, ο κύριος Κέλλη. Με κύριος ήμουν και τελευταία φορά που κοίταξα. Εμάς περιπτώσει με διαβεβαίωσε και η γυναίκα μου. Εντάξει, ναι, ναι, είμαστε βέβαιοι όλοι. Λοιπόν, ε, το... Ε, έχω το συνέστημα ότι αυτά τα έχουμε πει και ξαναπεί. Ε, τα έχουμε ξανασυζητήσει με τις σχετικές απόψεις οι οποίες ήταν παρεμφερείς. Οπότε, εάν θέλουμε κάποτε να φτάσουμε στο στόχο τον οποίον επιδιώκουμε, επιγόντως, με τόσες πολλές τροπολογίες από τις διάφορες επιτροπές ε, θα υπάρξει ένα διέξοδο. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να έχουμε και τις πληροφορίες ε, για τους καταναλωτές με μία εύκολη μορφή η οποία μπορεί να γίνει γρήγορα κατανοητή και να διασφαλίσουμε ότι η εσωτερική αγορά δεν θα επηρεαστεί. Αυτό είναι πολύ βασικό και μετά έχετε όλα τα τεχνικά θέματα. τα οποία μπορούμε να συζητάμε εσαΐ. Προσωπικά πιστεύω ότι το ινόπνευμα πρέπει να περιληφθεί. Δεν είμαι βέβαιος ότι θα μπορέσουμε αυτό το θέμα να το συζητήσουμε ε, χωριστά κάποια άλλη στιγμή. Και όσον αφορά το, τους κωδικούς με χρώματα, πρέπει να βρούμε μια συμβιβαστική λύση η οποία να βασίζεται στα χρώματα για να μπορέσουμε ε, να καταλήξουμε κάπου. Διότι αν δεν έχουμε ε, ε, κωδικούς με χρώματα, τότε ο στόχος του ότι προσπαθούμε να επιτύχουμε θα αποτύχει. Πρέπει λοιπόν να μην αφαιρέσουμε, να μην μειώσουμε τις επιλογές των ανθρώπων, να μην τους ε, επηρεάσουμε σε κάποια κατεύθυνση που δεν έχει σχέση με την υγεία τους και να βρούμε κάποιον άλλο τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουμε να έχουμε τις, ε, ε, τα χρώματα, όχι μόνο κόκκινο, ο, ε, μπέζ και πράσινο και πρέπει να δούμε ε, πόσο όλα αυτά θα διατυπωθούν για να είμαστε βέβαιοι ότι όλα αντιπροσωπεύονται, παρουσιάζονται σωστά και όλοι το γνωρίζουν. Θα πρέπει λοιπόν αυτό να το αποφασίσουμε. Οπότε αισθάνομαι ότι ε, δεν προχωράμε σωστά. Πηγαίνω σε μία λαϊκή αγορά όταν είμαι στο σπίτι, στην περιοχή μου και βεβαίως αυτού του είδους αγορές δεν πρέπει να υπόκεινται σε όλη αυτή τη ρύθμιση αλλά θα πρέπει να, να μην χρειάζεται ίσως να μας πούνε πόσο πόσα μήλα και ποιο ποσοστό είναι μήλα, πόσο ζάχαρη και ούτω καθεξής, αλλά τουλάχιστον να μας λέει ότι αυτή η τάρτα έχει μέσα α, μήλα, βούτυρο, ζάχαρη και ούτω καθεξής, για να μην επηρεαστούν ε, ε, υπερβολικά και πευλάς κόστους της σήμανσης. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας και κάτι τελευταία πράγματα. Σύμφωνο ότι πρέπει όλα αυτά να αρχίσουμε να τα χρησιμοποιούμε πολύ συγκεκριμένα ε, και νομίζω ότι αυτό είναι σαφές. Ε, Συμφωνώ ότι ε, ή θα υπάρχουν ή δεν θα υπάρχουν οι απαγορεύσεις. Είναι ένα θέμα που έχουμε ξαναεξετάσει. Εάν λοιπόν εξετάσουμε από διαφορετική οπτική γωνία τους στόχους που επιζητούμε να επιτύχουμε, θα πρέπει να υπάρξει και κάποια εκπαιδευτική προσπάθεια, διότι διαφορετικά θα έχουμε χάσει την ευκαιρία και πολύ χρόνο διότι η διαδικασία πρέπει να ξεκινήσει αμέσως και όχι μόνο αυτό, αλλά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα μπορέσει να είναι χρήσιμη. Και εάν αυτό δεν γίνει, νομίζω θα έχουμε χάσει μια εξαιρετική ευκαιρία. Ευχαριστώ. Τώρα δίνω το λόγο στον κύριο Γιούαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Άρα, ουσιαστικά συμφωνούμε όλοι ότι πρέπει να καθορίσουμε έναν γενικό στόχο για καλύτερη πληροφόρηση στον καταναλωτή. Επ' αυτού του θέματος συμφωνούμε. Το θέμα είναι να βρούμε την τεχνική με την οποία θα καταλήξουμε στην καλύτερη πληροφόρηση για να μπορεί να είναι ενημερωμένος και αναλόγως να επιλέξει. Ξέρετε που υπάρχει πιο αυστηρή νομοθεσία εκεί όπου είναι, υπάρχουν περισσότεροι παχύσαρκοι, δηλαδή στι Ηνωμένε Πολιτείες. Όταν λοιπόν τρώτε κάτι ε, πρέπει να πεινάτε πολύ διότι η σήμανση και η ετικέτα θα πρέπει να σας αποτρέψει και παρόλα αυτά 50% των ε, πολιτών είναι παχύσαρκοι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχει σήμανση, αλλά ίσως ε, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι δεν έχουμε βρει την ε, λύση του προβλήματος της διατροφής. Δηλαδή δεν θα καταφέρουμε ε, το στόχο, να επιτύχουμε το στόχο μας μόνο μέσω της σημάνσεως και επιπλέον πάρα πολλές πληροφορίες πάνω στην ετικέτα την ε, καταστρέφουν. Δηλαδή θα πρέπει ο πελάτης να καθίσει να αναλύσει όλα αυτά τα στοιχεία. Και από την άλλη πλευρά εμείς ε, υποκείμεθα στην πίεση ε, πολλών οι οποίοι θέλουν να ε, εγγράψουν τα προβλήματα που τους δημιουργούν προβλήματα. Δηλαδή οι διαβητικοί θέλουν να μιλάμε για τη ζάχαρη, η παχύσαρχη ε, για τα λιπίδια, η υπερτασική ε, για το αλάτι. Ο καθένας λοιπόν λέει τα δικά του. Πρέπει λοιπόν να μην τους δίνουμε μεγαλύτερες προσδοκίες από αυτές τις οποίες θα μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε ε, από πλευρά σήμανσης. Επιπλέον υπάρχει το θέμα των χρωμάτων, κόκκινο, κίτρινο και πράσινο τεχνικά. Εάν μιλούσαμε για κόκκινο, κίτρινο, πράσινο, θα έπρεπε να βάλουμε κόκκινο στην κοκακόλα. Ότι που σε, γρήγορη, ε, σε γρήγορα τρόφιμα όπως τα McDonald's, στι τηγανιτές πατάτες και είμαστε στο Βέλγιο. Ε, όταν μιλάμε δηλαδή για κόκκινο, ίσως κάποια μέρα θα ζητήσουμε να απαγορευτεί αυτό το τρόφιμο εφόσον είναι κόκκινο, δηλαδή ε, δεν πρέπει να καταναλώνεται. Τότε λοιπόν θα έπρεπε να έχουμε μία σήμανση που να μην είναι επιβαρημένη και να μην είναι ε, υπερβολικά απλοποιημένη σαν καρικατούρα με το κόκκινο, πράσινο κίτρινο. Ε, διότι ο καταναλωτής θα πρέπει να ενημερωθεί και να μπορέσει να τα βγάλει πέρα. Μετά, όσον αφορά τα μη προσυσκευασμένα τρόφιμα. Έχουμε ας πούμε την παγκέτα ψωμί στη Γαλλία και οι Γάλλοι ε, ε, παρουσιάζονται με ένα μπερεδάκι και ε, μία μπαγκέτα. Δεν μπορώ λοιπόν να πάω να πάρω μία μπαγκέτα η οποία θα έχει, θα έχει ιδιαίτερη συσκευασία για να μου αναφέρει τι περιέχει. Δεν είναι δυνατόν. Άρα όλα αυτά τα θέματα δεν μπορούν να υπόκεινται στην ε, ίδια νομοθεσία και θα πρέπει τα κράτη-μέλη να κρατήσουν για αυτούς τους τύπους προϊόντων. Δηλαδή ε, ε, τα μη συσκευασμένα ή τα συσκευασμένα ακριβώς πριν την πώληση τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τα θέματα ε, λαμβάνοντας ε, υπόψη τις ιδιομορφίες ε, και ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας. Επίσης, η μικρή παραγωγή ίσως θα πρέπει εν μέρη ή τελείως να εξαιρεθούν από αυτή τη ρύθμιση διότι δεν θέλουμε να αποδυναμώσουμε ε, το οικονομικό στοιχείο που συμβάλλει στον πλούτο της εσωτερικής αγοράς. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει η κυρία Γκέμπχαρτ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ αγαπητή Κρίστελ για την εργασία σου που είναι πραγματικά ιδιαίτερα σημαντική και καθόλου εύκολη και βασίζεται σε αυτό το οποίο έκανε ήδη η Μπερνατέτ στο παρελθόν. Και η συζήτηση σήμερα έδειξε πόσο δύσκολο και πολύπλοκο είναι το θέμα αυτό. Και θα πω ότι έχει δίκιο ο κ. Ζουβά που είπε ότι όλοι έχουμε τον ίδιο στόχο, δηλαδή να φροντίσουμε ούτως ώστε οι πολίτες να έχουν κάποια βοήθεια κατά την επιλογή σου, να έχουν αξιόπιστα δεδομένα που να μπορούν να βασιστούν σε αυτά. Ε, στη σύντηση αυτή θεωρώ ότι υπήρξε μια σύγχυση, δηλαδή συγκρίνονται τα μήλα με τα χλάδια. Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε λοιπόν περί τίνος συζητούμε εδώ. Εάν κατάλαβα σωστά και η Κρίστελ παρακαλείται να με διορθώσει αν κάνω λάθος, δεν συζητάμε για το χυμό μήλου γιατί νομίζω ότι είναι ε, αρκεί αν γράφει στην ετικέτα με προσθήκη ζάχαρης ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή δεν μιλάμε για το κομμάτι κρέας ε, ή τα λαχανικά στην ε, λαϊκή αγορά. Μιλούμε για συσκευασμένα τρόφιμα, ε, μείγματα τροφίμων, μικτά τρόφιμα μάλλον, όπου τα οποία είναι συσκευασμένα στην αγορά και όπου οι πολίτες δεν μπορούν να αξιολογήσουν περί τίνος ακριβώς πρόκειται, τι ακριβώς αγοράζουν. Εγώ πήγα στο σούπερ μάρκετ και προσπάθησα να δω διάφορα γλυκά. Ε, το γλυκό δεν είναι ωφέλιμο για την υγεία, εμένα μου αρέσουν όμως τα γλυκά. Ε, κοιτάω λοιπόν την περιεκτικότητα, κοίταξα λοιπόν την περιεκτικότητα σε λίπος και σε ζάχαρη κλπ. Και, και διαπίστωσα ότι δεν έχω καμία δυνατότητα σύγκρισης μεταξύ των διαφόρων προϊόντων. Γιατί ναι μεν αναφέρεται ε, αλεύρι, ζάχαρη κλπ. Τα συστατικά, αλλά δεν είναι δυνατή η σύγκριση μεταξύ των δύο προϊόντων. Δεν μπορώ να αποφασίσω τι είναι πιο ωφέλιμο μεταξύ δύο προϊόντων. Και νομίζω ότι αυτό είναι το ζητούμενο. Σε αυτή την ερώτηση θα πρέπει να δώσουμε μια απάντηση. Δίκαιο δεν έχω, κρίστερ. Ωραία. Το θέμα είναι πώς ε, μπορούμε να εξασφαλίσουμε τη συγκρισιμότητα. Η κυρία Ρούλα αναφέρθηκε στο τσάι για τα παιδιά. Και εδώ θα ήταν ε, σημαντικό. Ε, Ευτυχώ έχει καταργηθεί πλέον αυτό το τσάι. Να μπορεί να ε, γιατί παλιά το πουλούσαν χωρίς να αναφέρει την περιεκτικότητα σε ζάχαρη και αυτό είναι ιδιαίτερος επισήμιο για πολλά παιδιά. Θα έπρεπε λοιπόν να αναφέρεται στη συσκευασία η περιεκτικότητα σε ζάχαρη και θα έπρεπε να υπάρχει ένα κόκκινο σήμα που να λέει προσοχή ε, πόσο τσάι θέλετε να δώσετε στα παιδιά σας ή μήπως δεν θα πρέπει να προτιμήσετε ένα άλλο τσάι για τα παιδιά σας με χαμηλότερη περιεκτικότητα στη ζάχαρη. Και εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει μια μικρή διαφορά ε, όσον αφορά τη δική μου προσέγγιση για αυτή της κρίστελ. Δηλαδή, θεωρώ ότι δεν είναι χρήσιμο να έχουμε ένα σήμα ένα φανάρι ε, για το προϊόν, το ίδιο το προϊόν, αλλά για τα συστατικά του προϊόντος. Όχι κύριε Ζουβέ, δεν έχετε δίκιο. Στα προϊόντα αυτά έχουμε ήδη την περιεκτικότητα σε αλάτι, σε λιπίδια και λοιπά, σε ζάχαρη, λίπος και λοιπά. είναι υποχρεωτική αυτή η αναφορά. Ε, μπορεί αυτό να, γίνει, να τονιστεί με το χρώμα για τη ζάχαρη πράσινο και για το λίπος κόκκινο, δεν ξέρω, ανάλογα με τη σύνδεση του προϊόντος. Και το, στην περίπτωση αυτή ο πελάτης, ο διαβητικός, μπορεί να ξέρει ε, όταν δει το κόκκινο στη ζάχαρη ότι πρέπει να αποφύγει αυτό το προϊόν γιατί το θέμα δεν είναι η υγιής, το είπατε άλλωστε στο ίδιος. Υπάρχουν πολίτες που έχουν εντελώ διαφορετικές ε, παθήσεις και διαφορετικές ανάγκες σε ενημέρωση, σε πληροφορία και εμείς οφείλουμε να τους δώσουμε αυτές τις πληροφορίες για να μπορούν να πάρουν την κατάλληλη απόφαση όσον αφορά την υγεία τους. Και νομίζω <clears throat> ότι θα πρέπει να το διαμορφώσουμε έξυπνα. Να μην μπούμε ευθύ εξ αρχή αυτό το φανάρι κόκκινο, πορτοκαλί πράσινο είναι κακό, γιατί το κόκκινο σηματοδοτεί τον την απαγόρευση. Στο φανάρι σηματοδοτεί καταρχήν το ότι πρέπει να μείνουμε ακίνητοι, να μην περάσουμε και να δούμε κατά πόσο μπορούμε ή όχι να διασύσουμε τον δρόμο. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και όταν ε, δούμε ε, τη συζήτηση που γίνεται στις χώρες μέλη, βλέπουμε ότι οι πολίτες επιθυμούν ένα τέτοιο βοήθημα για να πάρουν ε, τις αποφάσεις αυτές, γιατί τα προϊόντα γίνονται όλο και πιο πολύπλοκα. Και αυτό είναι το θέμα εδώ γίνονται όλο και πιο πολύπλοκα τα προϊόντα, οι αποφάσεις γίνονται όλο και πιο δύσκολες σχέση με το τι μπορούμε να ψωνίσουμε και τι όχι. Δεν πρόκειται για το μήλο ή για το χυμό από μήλο, αλλά για τα πιο σύνθετα προϊόντα, τα fast food, τα οποία άλλωστε αναφέρατε κι εσείς. Αλλά στις Ηνωμένε Πολιτείε, η παχυσαρκία δεν ανάγεται στη σήμανση, αλλά σχετίζεται με το ότι δεν υπάρχει σωστή ενημέρωση. Για παράδειγμα, τα φυσικά προϊόντα. Ε, στα σούπερ μάρκετ στην Αμερική δεν υπάρχουν φρούτα ή λαχανικά. Αυτό είναι ένα εντελώς διαφορετικό πρόβλημα. Ε, και νομίζω θα πρέπει να το βάλουμε στην άκρη, γιατί οι αιτίε για τα προβλήματα στην Αμερική είναι εντελώς διαφορετικές στη Γαλλία, παρόλο που εκεί τα πράγματα επίσης αλλάζουν, είναι διαφορετική η κατάσταση. Γιατί εκεί στις αγορές υπάρχουν ε, πολλά μη συσκευασμένα φυσικά προϊόντα. Και εκεί δεν υπάρχει καμία ανάγκη σήμανσης. Αλλά ακριβώς εκεί που υπάρχουν οι συσκευασίες, εκεί υπάρχει ανάγκη. Παρακαλώ λοιπόν να μην ε, προκαλείται αυτή η σύγχυση και να μην δίνετε παράδειγμα τα οποία μας εκτροχιάζουν, μας ε, απομακρύνουν από το στόχο μας. Ε, ε, θα πρέπει να δώσουμε τη λύση για προϊόντα που χρίζουν αυτή της σήμανση. Σας ευχαριστώ πολύ. Δίνω τώρα το λόγο στην κυρία Βερνιό. Ευχαριστώ. Συμφωνούμε όλοι ότι βρισκόμαστε μέσα σε μια κοινωνία της αγοράς και έχουμε μάλιστα κάποια τύχη γι' αυτό, γιατί μπορούμε να επιλέξουμε, αλλά το να μπορούμε να επιλέξουμε και να μπορούμε να κάνουμε μια υπεύθυνη επιλογή, θα πρέπει βεβαίως να είμαστε καλά ενημερωμένοι. Και εγώ είμαι πεπισμένη και έχει γίνει μια πολύ τεχνική συζήτηση, όλοι συμφωνούμε επί του στόχου. Είναι αλήθεια, έχετε δίκιο ότι δεν είναι η ετικέτα, κύριε Ζουβέ, που θα βελτιώσει την υγεία εν μία νυχτή. Θα περάσουν χρόνια εκπαίδευσης στην υγεία και στην κατανάλωση. Δουλεύουμε για τις επόμενες γενναίες. Αυτό είναι το ευρωπαϊκό όραμα. Και εγώ πιστεύω σταθερά πώς μπορούμε να προσπαθήσουμε να συνοηθούμε. Αυτό υπάρχει ήδη για ορισμένα προϊόντα. Είχα αυτό το υπόθεση την τελευταία θητείας και πραγματικά εγώ τα βάζω τα γυαλιά μου όταν κάνω ψώνια. Υπάρχουν ένα σώρο προϊόντα, είτε είναι γαλακτοκομικά, είτε είναι έτοιμα προς κατανάλωση, υπάρχουν ήδη ετικέτες. Και τώρα για το φανάρι, για το κόκκινο, πράσινο κτλ. Υπάρχουν κάποια κατόβλια για πολλά θέματα και πρέπει αυτό ίσω να το σκεφτούμε. Πάντω υπάρχουν ήδη σημεία, υπάρχουν ήδη προϊόντα που ε, σηματοδοτούνται με διαφορετικά χρώματα. σω θα μπορούσαμε να συνεννοηθούμε στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Ένα Ούγγρο που έρχεται στη Γαλλία να καταλαβαίνει τα ίδια χρώματα, τα λιπίδια τάδε χρώμα, τα η ζάχαρη τέτοιο χρώμα και και ούτω καθεξής. Όταν βλέπουμε ότι ένα προϊόν περιέχει 75% λιπαρά και 30% ζάχαρη, να έχουμε την κατάλληλη παιδεία, ξέρουμε πως είναι επικίνδυνο αν το καταναλώνουμε τακτικά. Άρα λοιπόν μπορούμε να συμφωνήσουμε για μια απλή ετικέτα με χρώματα που θα αποδώσουμε σε κάθε κατηγορία, με μια καλή εκπαίδευση ε, αλλεργιογόνα, ζάχαρη και αλάτι. Γιατί συχνά τα αλλεργιογόνα αναφέρονται με κάτι μικροσκοπικά γράμματα και επειδή τα παιδιά και οι έφηβοι ε, έχουν την τάση να αγοράζουν ό,τι να είναι γιατί υπόκεινται στις εξατήσεις τις από την τηλεόραση, στην τηλεόραση, άρα λοιπόν πρέπει να μπορούμε να το δούμε να σημειώνεται μπροστά στο μπροστινό τμήμα γλουτένι, ένα σωρό πράγματα. Μπορεί να είναι σοβαρά τα πράγματα. Τώρα όμω, άμα έχουμε ένα πακέτο τσίχλες τέτοιο, όπου πρέπει όλα να τα βάλουμε μικροσκοπικά ή αν έχουμε μια μεγάλη συσκευασία, μπορούμε να βάλουμε κάποιες είναι τεχνικό το θέμα, αλλά θα το συμφωνήσουμε, θα τα βρούμε αφού συμφωνούμε επί του στόχου. Είχαμε σε αυτή την Επιτροπή Εσωτερική Αγορά κάνει μια ψηφοφορία που δεν ήταν και τόσο κακή. Πιστεύω πω θα πρέπει να επανέλθουμε και η πρόταση τη Κριστέλα νομίζω πω είναι λογική. Υπάρχουν ίσω κάποιε λεπτομέρειε που θα πρέπει να ρυθμίσουμε μεταξύ μα, αλλά νομίζω να είμαστε ενωμένοι σε αυτό το θέμα γιατί είναι ένα θέμα το οποίο φαίνεται να είναι ανώδυνο, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα, αν δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις, θα δώσω το λόγο στην ε, Κομισιόν. Δεν υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος εδώ. Ο κύριος Μαθιουδάκης. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Ήταν πολύ ενδιαφέρον να ακούσω τις ε, συζητήσεις, αλλά έχω ε, συγκρατήσει τα ουσιαστικά σημεία τα οποία παρουσιάστηκαν και ένα από αυτά ήταν ότι με αυτή την νομοθεσία θα δώσουμε τη δυνατότητα στον καταναλωτή να συμφωνήσει με την πρότασή μας. Δηλαδή να έχει πληροφόρηση ο καταναλωτής και να μπορεί να αποκομίζει πληροφορίες χωρίς ε, να χρειαστεί να ε, κάνει πάρα πολλές επιλογές. Η Επιτροπή βέβαια δεν θα πρέπει να υπερβάλλει γιατί η υπερβολική πληροφόρηση καταστρέφει την πληροφόρηση και γι' αυτό το λόγο προσπαθήσαμε να παρουσιάσουμε σε πολλά θέματα και τα στοιχεία τα οποία ε, ενδιαφέρουν τον καταναλωτή για να μπορέσουμε όλα αυτά να τα έχουμε σε μία θέση για να προσελκύσουμε την προσοχή του γιατί στο τέλος ο καταναλωτής δεν κοιτά την ε, ενημέρωση είτε γιατί δεν καταλαβαίνει όλα αυτά τα περίπλοκα είτε γιατί δεν τον ενδιαφέρουν πλέον. Ελέγχθη επίσης ότι θα έπρεπε ο κόσμος να μπορεί να κοιτάξει τις ε, ετικέτες και να τις διαβάσει με κανονικά γυαλιά. Με απλά γυαλιά. Και μετά από έρευνα διαπιστώσαμε ότι αυτός ήταν ένας βασικός λόγος για τον οποίο οι καταναλωτές δεν κοιτούσαν την πληροφόρηση διότι δεν ήταν εύκολο να τη διαβάσουν. Θέλω λοιπόν να πω στον κύριο Κρέχμαν ότι έχουμε προτίσει, προτείνει διάφορες λύσεις οι οποίες όμως δεν έχουν δεν έχουν βοηθήσει την πρότασή μας διότι είναι ο τρόπος με τον οποίο προχωρήσαμε. Μετά λοιπόν από συζητήσεις που έγιναν στο Συμβούλιο μπορούμε να πούμε ότι αυτό τώρα έχει διευκρινιστεί και συμφωνούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο μέγεθος όπου θα προβλέπετε ότι πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον το τάδε ε, μέγεθος ε, γραμμάτων και ότι θα πρέπει να καλύπτουν δύο χιλιοστά από 2,5 που έλεγε αρχικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτά μπορούμε να τα υιοθετήσουμε εφόσον τα έχει δεχθεί και το Συμβούλιο. Και τέλος, ακούσαμε πολλά σχετικά με τις ε, προτιμήσεις των μεν, προτιμήσεις των ε, άλλων, ε, δηλαδή κωδικούς χρωμάτων, οι GDAs που μπορούν να βοηθήσουν τον καταναλωτή να αξιολογήσει τον αριθμό των θερμίδων τις οποίες προσλαμβάνει. Άκουσα όμως ότι ελπίζουμε ότι θα υπάρξει νομοθεσία η οποία θα είναι χρήσιμη σε επόμενες γενιές. Οπότε μαζί με τις διατροφικές πληροφορίες ελπίζω ότι θα υπάρξουν και τα στοιχεία αυτά αλλά όσον αφορά τα σύμβολα και ε, τους κωδικούς χρωμάτων πιστεύω ότι σήμερα δεν έχουμε επαρκείς πληροφορίες για να μπορέσουμε να επιβάλλουμε ένα σύστημα. Γι' αυτό και πιστεύουμε ότι η ιδέα του να επιτρέψουμε να αναπτυχθούν προγράμματα συμβουλευτικά που, στα οποία θα εμπλακούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι και όπου θα υπάρχει και κάποια εποπτεία των ε, κρατών ε, μελών, δηλαδή όχι επιβολή αλλά εποπτεία των κρατών μελών κατά τρόπον ώστε να αναπτυχθούν συστήματα τα οποία θα μπορέσουν να εφαρμοστούν και όταν θεωρήσουμε ότι ένα από αυτά τα συστήματα έχει γίνει ε, κατανοητό από όλους τους πολίτες στην κοινότητα τότε θα μπορέσουμε να εναρμονίσουμε ε, τα προγράμματα διότι τα εθνικά προγράμματα δεν θα αποτελέσουν και τέτοιο πρόσκομα ακούσαμε ότι αν επιτρέψουμε εθνικά προγράμματα ε, θα έχουμε 25 συστήματα τα οποία θα πρέπει να πολλαπλασιαστούν στις εταιρείες αλλά οι εταιρείες ε, ε, είναι πολυεθνικές και τελικά θα υπάρξει ένα μόνο πρόγραμμα και θα μπορέσουμε να προτείνουμε διάφορα θέματα για να τα έχουμε ε, κατά τρόπον ώστε να μην ε, ε, μας ενοχλήσουν. Main voluntary schemes. Διότι υπερβολικά πολλά προγράμματα νομίζω θα κατακαιρματίσουν τις αγορές. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω και Ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να παρουσιάσω την πρόταση αυτή, διότι ε, έχει μεγάλη σημασία και πολλές επιπτώσεις και φαντάζομαι ότι θα πρέπει να αξιολογηθεί ιδιαιτέρως. Io la ringrazio per il eh, suo contributo e eh, ritengo che sia stato assolutamente puntuale. Ευχαριστώ ε, γιατί ήσασταν ακριβείς ε, και δώσατε χρήσιμες πληροφορίες που θα χρησιμεύσουν στους εισηγητές και στους σκιώδεις. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Σαλδεμόζερ η οποία θα ε, καταλήξει και θα παρουσιάσει τα συμπεράσματά της. Σας ευχαριστώ και σας ευχαριστώ για όλα αυτά τα εξαίρετα σχόλια. Θα ε, ε, εκτιμώ ότι είχαμε περισσότερο χρόνο για τη συζήτηση, γιατί πολλοί ήθελαν να συμμετάσχουν. Θα ήθελα να κάνω μερικά σχόλια και να αφήσω τη συζήτηση για το μέλλον. Όταν μιλάμε για μια κομμεδικοποίηση μέσω χρωμάτων, για αυτά τα φανάρια της κυκλοφορίας, όπως θέλετε να το αποκαλέσετε, θα πρέπει να αποφασίσουμε πώς θα το κάνουμε. Ή θα, αν θα αναφέρονται στα συστατικά ή τα ποσοστά κλπ. Νομίζω ότι αυτό δεν παίζει τόσο ρόλο. Σημαντικό είναι να δώσουμε στον καταναλωτή τη δυνατότητα να κατανοεί τι περιλαμβάνει